Sorry, Πρέπει να αρχίσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι η Μόνικα Χολμαϊρ που είναι η συγγήτρια για το σημείο 4 δεν έχει έρθει ακόμα. Αν κάποιο έχει το τηλέφωνο τη να την ενημερώσει, μπορούμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη. Θα πρότεινα όμως να αρχίσουμε με τηρώντα την ημερήσια διάταξη μια και είναι πρώτη μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Να σας καλωσορίσω όλους και τη Μόνικα. Καλώς Η συγγήτρια που περιμέναμε. Καλώς ήλθατε όλοι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Και τώρα θα αρχίσουμε την πρώτη συνεδρίασή μας. Ημερήσια διάταξη Εναν σας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τότε υιοθετείτε. Ελπίζω να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Έχεις ακόμα λίγο χρόνο, Μόνικα. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Και έχουμε δύο πρακτικά, δύο συνεδριάσεων, της 12ης Ιανουαρίου και της 12ης Απριλίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, τότε τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Τώρα, ας αρχίσουμε με το σημείο 4, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020 και η συγγήτριά μας Μόνικα Χολμάιερ αυτή τη στιγμή ψάχνει τα χαρτιά της. θα συζητήσουμε τις τροπολογίες, το σχέδιο γνωμοδότησης του, δημοσιο... του δημοσιονομικού πλαισίου και αν η Μόνικα είναι έτοιμη τότε με χαρά θα της δώσω το λόγο. Και μετά θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη, εάν επιθυμούν, να πάρουν το λόγο και να παρέμβουν. Μόνικα, παρακαλώ. Δώσε μας την Πρέληψή σου. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μόλις τώρα ήρθα από άλλη συνεδρίαση, γι' αυτό σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε για την ε, μικρή εργοπορία μου. Ε, τώρα έχουμε να κάνουμε με την γνωμοδότησή μας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που ε, ήταν συνεισηγητές και εσείς κύριε Πρόεδρε ήσασταν μαζί που συνεργαστήκαμε. Τώρα όσον αφορά τα σημεία που ήθελα εγώ να τονίσω στις προτάσεις μου, αυτά θα σας παρουσιάσω. Καταρχάς, ε, συνειδητοποίησα ότι το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και η χρηματοδοτική δομή του χρήζει απλούστευσης, ακριβώς όπως και το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια και την εισαγωγή ε, ενιών προδιαγραφών για την δίκηση, τον έλεγχο και την ε, υποβολή αναφορών. Επιπλέον, έχω κάποιες ε, αμφιβολίες για το, αν για το ότι η χρηματοδότηση για τα προγράμματα, δεν θα είναι και τόσο εύκολη για τα προγράμματα στους τομείς που μας αφορούν επιπλέον. Συζητήσαμε μεταξύ μας για, τα, για τις ε, ε, εργασίες που πρέπει να κάνουμε και να διαπραγματευτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχίζουμε με το κυβερνοέγκλημα, με, το σύμφωνο για τα, τα PNR των επιβατών, για το άσυλο, Συνειδητοποίησαμε λοιπόν ότι η χρηματοδότηση είναι σχεδόν ανεπαρκής. Έχουμε κάποιες τροπολογίες από τους αγαπητούς συναδέλφους. Ε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις επικοδομητικές συνεισφορές τους. Ε, συζήτησα ε, και με τους συναδέλφους συμφωνήσαμε για να συμβιβαστούμε σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα για ένα συνετό χρηματοδοτικό όργανο για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. στο τομέα της ασφάλειας, της ελευθερίας και του δικαίου στο πολιετές δημοσιονομικό πνέσιο. Για παράδειγμα, η πρόεδρος κυρία Βίκστρομ, οι συνάδελφοι Τόμσον συνείσφεραν για τους ε, τομείς ε, δικαιώματα και ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ε, καταλήξαμε σε μία ε, καλή κοινή θέση. Υπήρξαν προσθήκες από τον συνάδελφο Γκιόμ όσον αφορά το, άσυλ, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και τέλος θα προσπαθήσω μαζί με όλους εσάς να καταλήξουμε σε μία πρόταση όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής στις ε, προσεχείς ημέρες θα συνομιλήσω με, τους, ε, με τον συνάδελφο Χάλτεν, ε, με τους συναδέλφους μου μάλλον και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να σας επαναλάβω τα επιμέρους σημεία των τροπολογιών Έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι οι 16 που έχουμε εδώ είναι αρκετές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την περίληψη. Εντάξει, οι τροπολογίες είναι καλός αριθμός. Οι 16 τροπολογίες είναι καλές. Η κυρία Κέλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα προσθέσω πάρα πολλά. Θα ήθελα να συμμετέχω στη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την δουλειά και με πολύ χαρά είδα ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους τόνισαν την σημασία της προστιθέμενης αξίας στα προγράμματα δράσης μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίση θα ήθελα να υπογραμμίσω και να σα υπενθυμίσω το σύστημα τη αξιολόγηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τι σωστέ ε, αποφάσει όσον αφορά την χάραξη πολιτική. Ε, και αυτό θα το συζητήσουμε στην ψηφοφορία για το προπολογισμό του 2013 βέβαια στη συνέχεια. Α έχουμε όμω υπόψη ότι οι αξιολογήσει είναι πολύ σημαντικέ για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλοι πρόεδρο. Και εγώ θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα ως ε, συνεισηγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χολμάιερ για την δουλειά σας. Από τη μία έχετε δίκιο, ε, οι 16 τροπολογίες είναι κάτι από το από την άλλη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με το σύνολο των ε, λεπτομεριών του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου. Ζητούμε όμως και ισορροπία σε αυτό και οι τροπολογίες που καταθέσαμε ε, λίγο πολύ προσπαθούν να επιτύχουν αυτήν την ισορροπία που επιθυμούμε στην ε, κατανομή των κονδυλίων τα οποία πρέπει να συναδούν με τις ενές δομές ε, την απλούστευση την συνέχιση, την ομαλή συνέχεια των προγραμμάτων και αυτών των ε, οργανισμών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει προβλεψιμότητα, να ξέρουμε τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Να δούμε ποιοι είναι οι σημαντικότεροι στόχοι μας και να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι αυτοί θα, θα καλυφθούν από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ακόμα και αν χρειαστεί να συζητούμε κάθε χρόνο για τον προπολογισμό. Κάθε χρόνο ξεχωριστά. Οι τροπολογίε λοιπόν λίγο πολύ ασχολούνται με αυτό το θέμα και από όσο βλέπω δεν υπάρχουν σοβαρέ διαφωνίε. Μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ τροπολογίε και να οδηγηθούμε σε μια ψηφοφορία που θα δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτό θα ήθελα να δω μέχρι το τέλος. Κύριε Μπρόνξ, θα θέλετε να πάρετε το λόγο. Μάλιστα. Η κυρία Χολμάιρ έχει προφανώς δίκιο για το ότι το πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη τις αυξανόμενες υποχρεώσεις στην, ε, στο, στον τομέα της ελευθερίας, του δικαίου και της ασφάλειας. Ανέφερε την ίδρυση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης και την τροποποιημένη εντολή του Frontex. Εάν τα κονδύλια είναι ανεπαρκή, μπορούμε είτε να δούμε τα κονδύλια, είτε να δούμε τις ε, αρμοδιότητες. Προτείνω να δούμε τις αρμοδιότητες και να αντικατασταθεί το Ταμείο Σύλλου και Μετανάστευσης με ένα άλλο Ταμείο της Πρόληψης. Έπειτα, η Frontex χρειάζεται καινούργια εντολή, βέβαια, έτσι ώστε να μπορεί να κρατεί τους ετούντες άσυλο και τους παράνομους μετανάστες μέχρι ότου να μπορέσουν να επιστραφούν στις χώρες τους. Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει φυσικά εντός ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση ανθρώπων που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα, τότε είναι σημαντική η έγκαιρη επιστροφή τους και η ανάγκη για τα κονδύλια θα μειωθεί αν διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μούλτερ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε κάτι ε, για το στο οποίο δεν αναφερθήκαμε και δεν ξέρω αν έχει συνυπολογιστεί ή όχι και που αφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση περισσότερο είναι το γεγονός ότι εξοικονομούμε χρήματα για τα κράτη-μέλη διότι ο συντονισμός που κάνουμε δεν γίνεται ε, ως εκ τούτου μεμονωμένα από κάθε κράτος μέλος. Στου επόμενου μήνε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ίσω κάποιο από την Επιτροπή, από τη Γραμματεία τη Επιτροπή μα ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να έχει κάποια στατιστικά στοιχεία για την εξοικονόμηση πόρων ε, για τα κράτη-μέλη. Αν αναλάβουμε εμεί κάτι σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αυτό θα βοηθούσε. Ε, είναι προφανέ ότι έχουμε έλλειψη πόρων και όλοι θέλουν να περιστύλουν τι ε, δαπάνε του. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε, με, ε, υποστηρίζοντας το με συγκεκριμένα στοιχεία, ότι εξοικονομούν χρήματα τα κράτη-μέλη. Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ. Η κυρία Καριγιό είναι εδώ εκπροσωπώντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να μας απαντήσετε. Να μας πείτε αν έχετε στοιχεία αριθμητικά για την εξοικονόμηση πόρων ή αν θα συζητηθεί καν αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για ποιο λόγο δηλαδή είναι πιο συνιστά καλύτερη χρήση των πόρων το να ε, κινούμεθα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξοικονομώντας ε, χρήματα από τον εθνικό συντονισμό. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, Μόνικα, ζητάει το λόγο. Ενδεχομένως να δώσουμε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει ή όποιος ε, άλλος το επιθυμεί, ο πλευράς του Συμβουλίου και στη συνέχεια να σας ακούσουμε. Η κυρία Καριγιό από πλευράς Επιτροπής. Ε, αν έχετε μία απάντηση λοιπόν για αυτή την ερώτηση ή οποιαδήποτε άλλα σχόλια σας ακούμε. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω συγκεκριμένες απαντήσεις ε, τώρα. Αλλά πράγματι ο... οι προτάσεις ε, της Κομισιόν λαμβάνουν υπόψη την προστιθέμενη αξία του στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό πράγμα το οποίο δεν ε, αποτελεί οικονομία για τα κράτη-μέλη, αλλά λαμβάνουμε υπόψη μας τη δυνατότητα του να ξοδεύουμε με καλύτερο τρόπο συλλογικά, διότι ακριβώς υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη όσον αφορά στην καταμερισμένη ε, διαχείριση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οικονομία. Εδώ πρόκειται για αλληλεγγύη ε, πρόκειται για δράσεις οι οποίες είναι εθνικές ε, δράσεις, ε, οι οποίες θα είναι καλύτερης ποιότητας όταν είναι καλύτερα συντονισμένες, και υπάρχει μια καλύτερη έννοια, μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ διαχείρισης και αλληλεγγύης όταν έχουμε κοινέ δράσεις οι οποίες ε, δύσκολα μπορούν να αναλυφθούν από ένα και μόνο κράτος ε, μέλος. Εγώ σας ε, παραπέμπω, εάν θέλετε να δείτε καλύτερα τις οικονομικές επιπτώσεις, την μελέτη επιπτώσεων των προτάσεων της Κομισιόν αλλά όσον αφορά στο Ταμείο για τους ε, μετανάστες και για την εσωτερική ασφάλεια, εμείς εξετάσαμε από κοντά το θέμα της, ε, την έννοια της προστιθέμενης αξίας πριν υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Πρόκειται για μια ευρύτερη αντίληψη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και όχι οικονομίας. Ευχαριστώ. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι το ζητούμενο ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Μόνικα, παρακαλώ συνοψίστε τη συζήτηση μέχρι στιγμής. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να αναφερθώ ξανά στο ζήτημα της χρηματοδότησης των οικονομικών στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Πρέπει να βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, στο κυβερνοέγκλημα στον Ευρωπαϊκό Συντονισμό για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που, ε, για το οποίο έχουμε και ειδική υποεπιτροπή. Ε, χρειάζεται συνεργασία, γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν το καθένα μόνο του. Χρειάζονται συνεργασία, από κοινού αντιμετώπιση. Αγαπητέ συνάδελφε Μπρόνξ... Εάν δεν επενδυθούν χρήματα σε αυτούς τους τομείς, οι ζημίες θα είναι τόσο μεγάλες που πραγματικά είναι πολύ ωφέλιμο να δοθούν αυτά τα κονδύλια στον τομέα της ασφάλειας. Όσον αφορά το άσυλο και την ανθρωπιστική βοήθεια για τη μετανάστευση, ε, οφείλουμε να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη ή εκείνους στους οποίου, εκείνα τα κρατημέλη τα οποία δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να ε, καταρτήσουν ένα σύστημα ασύλου που να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο ευρωπαϊκός χώρος. Όσον αφορά την πρόταση της κυρίας Κέλλερ και του συναδέλφου Γκυγιόμ, συναδελφοί αυτοί ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το ζήτημα τη προστιθέμενης αξίας, όπως και εσείς, κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε τα χρήματα που θα επενδυθούν στην Ευρώπη να μην είναι αντικατάσταση εθνικών κονδυλίων, αλλά προσθήκη στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα, λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να έχουν μια πρόσθετη χρήση. Η κατανομή φυσικά των πόρων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ε, συνετότερη και κάποια έργα φυσικά έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από κάποια άλλα. Πρέπει να τεθούν αυτές οι προτεραιότητες. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα ε, να συνοψίσω με αυτά τα λόγια και ελπίζω να καταλήξουμε σε επικοδομητικές εργασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μόνικα είπε ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 19 και 20 του μήνα, στην επόμενη συνεδρίαση. Και τον Οκτώβριο έχει προβλεφθεί η συζήτηση για την, η ψηφοφορία συγγνώμη, για τον προϋπολογισμό. Έχουμε χρόνο δηλαδή για να τα ξαναπούμε και με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι το Eurodac. Η Μόνικα Μακκόβε είναι η συγγήτριά μας. Είχαμε προγραμματίσει την έναρξη για τις 3.30, ε, άρα υπολείπονται 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια νέα για τη Μόνικα, αν έρχεται, αν ε, πρέπει να, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ίσως μέχρι τις 3.30 δεν τη βλέπω τη Μόνικα εδώ μέσα. Διακόπτουμε. Διακόπτουμε για 10 λεπτά και αν στο μεταξύ μπορεί κάποιος να μάθει αν είναι καθοδόν ή όχι η Μόνικα, δεν έχει καταφτάσει. Λοιπόν, και 40 ε, θα ξεκινήσουμε και πάλι. 3 και 40.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 Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Ας ξαναρχίσουμε τη δουλειά. Να σας πω ότι η Επιτροπή ομόρφινε μετά τις θερινές διακοπές και να ζητήσω ξανά συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καθυστέρησε η από τη Μαδρίτη στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο που με αντικατέστησε στη σημερινή απογευματινή συνεδρίαση και συνεχίζουμε μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα με το σημείο 5 για την θέσπιση του Eurodac για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων, την αναδιατύπωση. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφός μας, κυρία Μακοβέη. Η πρόταση είναι ένα από τα μέτρα που χρειάζονται για την θέσπιση κοινού συστήματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναδιατύπωση του ισχύοντος κανονισμού από το 2000 και θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της Eurodac και περιέχει την δυνατότητα των αρχών επιβολής νόμου των κρατών μελών να συμβουλεύονται τα δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία έχουν επεξεργαστεί από την κεντρική βάση δεδομένων της Eurodac για τον σκοπό ε, ασκήσεως των καθηκόντων τους. Αυτή η πρόταση τροποποιεί την πρόταση της Κομισιόν του, ε, τον κανονισμό του 2000 που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η έκθεση συντάχθηκε από την συνάδελφο Μακοβέη και έλαβε υπόψη την ε, συνθήκη της Λισαβόνας στο μεσοδιάστημα. Τώρα λοιπόν, για να δώσουμε μία αγώνιμη βάση για συζήτηση, θα πρότεινα να ακούσουμε αρχικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα μας παρουσιάσει την τροποποιημένη πρόταση. Έπειτα να ακούσουμε την Κυπριακή Προεδρία και τέλος από την εισηγήτρια κυρία Μακοβέη. Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα, γι' αυτό να έχετε υπόψη την, το χρόνο που έχουμε. Ο λόγος περνά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. τον κύριο Ματίας Όιλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο φάκελος που συζητείτε σήμερα δεν είναι νέος, όπως είπατε. Το αντίθετο, από το 2008 και μετά έχει ένα μακρύ ιστορικό. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια παρουσίαση σε δύο μέρη. Πρώτον, να κάνω μια επισκόπηση των τελευταίων τεσσάρων ετών για το φάκελο Γιουροντά και να περάσω στη συνέχεια στην αναχείρας πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τον Ιανουάριο του 2003 και μετά λειτουργεί αισίως ε, το σύστημα Eurodac. Είναι μια πραγματική επιτυχία στον τομέα αυτό και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Όμως, το 2008 και βάσει τη αξιολόγηση ε, Δουβλίνο Eurodac πρώτη φορά πρότεινε κάποιε τροποποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προς το πεδίο εφαρμογή του Eurodac μέσω από σχέδια αναθεωρημένου κανονισμού και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για αυτό το θέμα το Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να επεκτείνουν περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου. Στην μία ανακοίνωση του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη αναφέρει ότι θα ήταν πρόσφορο κατά τη δική της άποψη να χορηγηθεί πρόσβαση για λόγους επιβολής του νόμου στο σύστημα Eurodac. Μετά το 2009 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή δύο νέοι κανονισμοί Eurodac, φάση πρόλης αβώνας, ε, εφόσον πρόκειτο για διαφορετικό πυλώνα και προτείναμε πρόταση, απόφαση Συμβουλίου για την πρόσβαση για την επιβολή του νόμου και υπήρχε ταυτόχρονα και ο κανονισμός Eurodac με bridging clause, μια ρήτρα δηλαδή που γεφυρώνει ε, του, τα δύο νομοθετήματα ως προς την πρόσβαση για τους λόγους επιβολής του νόμου. Στη συνέχεια τέθησε ισχύ η συνθήκη Λισαβόνας, καταργήθηκε αυτή η διάκριση των δύο πυλών και φτάνουμε έτσι στο 2010 όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλοντας να μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθεί το πακέτο το ασύλου μέχρι τα τέλη του 2012 κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρίτη και νέα πρόταση για το Eurodac που δεν, το τονίζω δεν, συμπεριλάμβανε την πρόσβαση για σκοπούς υποβολή νόμου. Κατά τη διάρκεια όλων των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο προέκυψε με σαφήνεια ότι τα κράτη-μέλη είναι μάλλον απρόθυμα να διαπραγματευτούν καλή την πίστη για το υπόλοιπο του πακέτου Eurodac ε, δίχως να συζητείται το θέμα τη πρόσβαση στα στοιχεία. Χάρη στην ε, αξιοσημείωτη πρόοδο που σημειώθηκε ω προ το πακέτο ασύλου κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντο έτου, Η επίτροπο ε, Μάλστρομ έκρινε ότι ήρθε η σωστή στιγμή η, απο... η νέα πρόταση για το Eurodac να συμπεριλαμβάνει ε, την επίμαχη διάταξη για την πρόσβαση στα στοιχεία. Αυτά ω προ το ιστορικό για να έχετε μια πλήρη εικόνα για τα τεκτενόμενα και θα περάσω τώρα στην ε, ουσία της πρότασης που εξετάζουμε σήμερα. Όπως ήδη είπατε, Πρόεδρε, πρόκειται για συγχώνευση ε, του νομοθετήμα το 2009 με ε, το Omnitext του 2010. Η διατύπωση ως εκ τούτου δεν έχει τροποποιηθεί ε, σημαντικά. Πρόκειται πραγματικά για συγχώνευση των δύο νομοθετημάτων. Το επεξηγηματικό σημείο που συνδέεται με την πρότασή μας στο τμήμα 7 αναφέρεται συγκεκριμένα στα άρθρα στα οποία, τα οποία προέρχονται από προηγούμενα σχέδια και τονίζει ποια είναι τα ε, νέα σημεία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να παρακολουθήσετε έτσι το φάκελο και να γνωρίζετε τι ε, ήδη ισχύει και τι νέο προτείνουμε. Όπω και στην πρόταση του 2009 και με τη νέα πρόταση, οι αρχέ επιβολή του νόμου θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να βλέπουν τα δακτυλικά αποτυπώματα που θα προμηθεύονται από τη βάση δεδομένων Eurodac μόνο υπό ε, αυστηρά προσδιορισμένε ε, περιστάσει και συνθήκε. Δεν Υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μας σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων, ούτε δρούμε κατά των συμφερόντων των ετούντων άσυλο ε, ή των μεταναστών με τη νέα αυτή διάταξη και θεωρούμε ότι επιτύχαμε μια πολύ ικανοποιητική ισορροπία με τη νέα πρόταση. Γιατί προτείνουμε λοιπόν πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac για τις αρχές επιβολής του νόμου. Είναι απλή η απάντηση. Θέλουμε να καλύψουμε ένα χάσμα, ένα κενό που υπάρχει θα σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.

Αυτή τη στιγμή, αν η αστυνομία κυνηγάει ένα δολοφόνο, μπορεί να συμβουλεύεται την εθνική βάση δεδομένων, ε, τη βάση δεδομένων που έχουν για τις εθνικές ταυτότητες, τις βάση δεδομένων άλλων κρατών μελών ε, ή τη βάση δεδομένων ε, του συστήματος ενημέρωσης για τις θεωρήσεις, για να καλύψει και τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ζητήσει θεώρηση, όμως δεν έχει δυνατότητα πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac. Και γι' αυτό σας είπα ότι καλύπτουμε ένα κενό που υπάρχει ε, δεν πλήττουμε καμία ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα και εξασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση αυτή είναι για την αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών και σοβαρών αξιοπίνων πράξεων. Μόνο και για αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η πρόσβαση. Είναι ένα ιδιαίτερα ακαθόδες και επίμαχο το ζήτημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ρήτρα διασφάλισης για να μην γίνει κατάχρηση της πρόσβασης σε αυτή τη χρήση δεδομένων. Άλλο ένα συγκεκριμένο και σύντομο παράδειγμα μια τέτοια ρήτρα διασφάλισης λοιπόν. Πρώτον, ε, καλύπτουμε την βάση επικουρικότητας μέσα στην πρόταση. Τι σημαίνει αυτό. Είναι η τελευταία, ε, το, η έσχατη λύση η πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Μόνο αν δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα από τη χρήση άλλων βάσεων δεδομένων, μπορεί κάποιο ε, να συμβουλευτεί τη βάση Eurodac. Τα κράτη-μέλη πρώτα θα συμβουλευτούν τα δακτυλικά αποτυπω... τις δικές τους βάσεις δεδομένων για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Στη συνέχεια θα κάνουν διασταυρωμένο έλεγχο με τις βάσεις δεδομένων άλλων κρατών μελών πάλι για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αν αυτές οι δύο έρευνες δεν καρποφορήσουν, τότε μόνο δικαιούνται να κάνουν μια επαλήθευση χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων Eurodac. Δεύτερον, η επαλήθευση γίνεται μόνο για σοβαρά εγκλήματα και τρομοκρατικές ενέργειες, όπως προσδιορίζεται αυτό από την απόφαση πλαίσια του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ξεκαθαρίσαμε ότι οι συστηματικές επαληθεύσει δεν επιτρέπονται. Επίσης, ξεκαθαρίσαμε ξεκαθαρίσαμε ότι η επαλήθευση για δακτυλικά αποτυπώματα για άλλες εγκληματικές ενέργειες επίσης ε, απαγορεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ρήτρα διασφάλισης προ τη χρήση. Ε, τώρα, όταν γίνεται μια επαλήθευση, το αποτέλεσμα θα δείχνει μόνο αν ένα κράτος μέλος έχει δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία για αυτό το έγκλημα. Τίποτα παραπάνω. Εάν ε, ε, ε, ζητείται επεξεργασία περαιτέρω προσωπικών στοιχείων, αυτό δεν καλύπτεται από την ελόγω διάταξη. Δηλαδή, εάν ένα δακτυλικό αποτύπωμα σε μια σκηνή εγκλήματο ταιριάζει με το δακτυλικό αποτύπωμα τη βάση δεδομένων Eurodac, τότε μόνο μπορεί να ζητήσει κανεί πρόσβαση για την επεξεργασία των στοιχείων. Κατόπιν δεν θα υπάρξει ανταλλαγή στοιχείων με τρίτε χώρε. Όλα αυτά τα στοιχεία θα παραμένουν στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εν κατακλείδη, Πρόεδρε, θα λέγαμε ότι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προχωρήσουμε ταχύτατα με το φάκελο Eurodac στα πλαίσια ε, της διαμόρφωσης ε, του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Θεωρούμε ότι είναι εξισορροπημένη η πρότασή μα ε, για την χορήγηση πρόσβαση στη βάση δεδομένων γυρώντα γιατί καλύπτουμε ένα προϋπάρχον κενό ε, συμπεριλαμβάνοντα απαιτούμενε ε, ρήτρε διασφάλιση, επικουρικότητα, δηλαδή περιορισμό στι τρομοκρατικέ ενέργειε και τα σοβαρά εγκλήματα, μη ανταλλαγή στοιχείων με τρίτε χώρε. Όλα αυτά τα στοιχεία ενσωματώνονται στο συνολικό ε, σύστημα σύλλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευελπιστούμε μέχρι το τέλο ε, του τρέχοντο έτου, να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για το συνολικό πακέτο θα ήθελα να το έχετε κατά νου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, διότι θα ήταν πλέον ατυχές να μην τηρήσουμε την καταληκτική ημερομηνία αυτή, δηλαδή το τέλος του 2012 για το συνολικό πακέτο ασύλου, μόνο και μόνο επειδή εκκρεμεί ο φάκελος Eurodac. Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κυπριακή Προεδρία που σήμερα εκπροσωπείται εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε προς το Συμβούλιο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούν και να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι κίνητρες διασφάλισης, στις οποίες προαναφέρθηκα και προσφέρουμε ε, την ε, συνεργασία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Ευχαριστούμε Πρόεδρο. Σας ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας τώρα. Ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου είναι το όνομα που μας έχουν δώσει. Παρακαλώ. ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας ενώπιον της Επιτροπής Δημοσίου Ελευθερών του Κοινοβουλίου. Όπως ήδη ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σχέδιο κανονισμού που εξετάζεται σήμερα είναι ένα σχέδιο το οποίο τα κράτη-μέλη ζητούσαν για αρκετό χρόνο, για, αρκετό για αρκετά μεγάλο διάστημα. Είναι ένα σημαντικό κείμενο για την ολοκλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και η, Προεδρία, η Κυπριακή Προεδρία ανέλαβε την εξέταση του θέματος ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω για την πορεία της εξέτασης του σχεδίου κανονισμού. Ήδη το σχέδιο εξετάστηκε δύο φορές στα πλαίσια της ομάδας εργασίας. Μια τρίτη συνεδρίαση της αρμόδιας ομάδας εργασίας είναι αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη και η φιλοδοξία και ο στόχος της Προεδρίας είναι να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Συμβουλίου το συντομότερο δυνατό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου μέσα στον επόμενο μήνα, κάτι που εξαρτάται προφανώς και από την πορεία των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την ε, Προεδρία και για τα κράτη-μέλη ε, το σχέδιο κανονισμού ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο Θεωρούμε ότι ε, ο κανονισμός Eurodac όπως λειτουργήσε μέχρι τώρα ήταν ένα χρήσιμο, εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός ε, Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον ε, με τις τροποποιήσεις που έχει επιφέρει η Επιτροπή θα αποτελέσει επίσης ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Όπως ανέφερε για τα κράτη-μέλη η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στις διοκτικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου είναι κάτι θετικό, ιδίως στο μέτρο που δεν ε, παραβιάζει δικαιώματα των ε, ετούντων άσυλο ή των ετούντων διεθνή προστασία και όπως ανέφερε και η Επιτροπή υπάρχουν σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες ε, τα κράτη-μέλη οφείλουν να τηρούν και αυτό είναι κάτι που ήδη στο Συμβούλιο δεν αμφισβητείται. Ευελπιστούμε λοιπόν για να κλείσω στην ολοκλήρωση της συζήτησης για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο ε, το συντομότερο δυνατόν μέσα στο Σεπτέμβριο αν γίνεται και περιμένουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο στην ε, διαμόρφωση της κοινή μας θέσης έγκαιρα ούτως ώστε να τιμήσουμε και να τηρήσουμε την προθεσμία του τέλους του 2012 για την ε, υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Now, we're ready to hear from... Σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα την εισηγήτριά μας, την κυρία Μακοβέη. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους ε, σκιώδεις η κυρία Μακόβε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που επέστρεψαν όλοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πολύ καλή περιγραφή του σχεδίου. Δεν χρειάζεται να επανέλθω. Καλωσορίζω λοιπόν τη νέα πρόταση Χαίρομαι που έχουμε αυτή την προσέγγιση, θετική ανταπόκριση ή όχι, χ, την hit. αυτή την προσέγγιση λοιπόν για την πρόσβαση, για τις αρχές επιβολής νόμου. Θα σπεύσουμε για να ολοκληρωθεί το αχύτερο δυνατόν η διαδικασία. Χαιρόμαστε επίσης διότι υπάρχουν ρήτρες διασφάλισης. Ε, προβλέπεται για τα κράτη-μέλη να συμβολεύονται πρώτα την εθνική βάση συνέχεια πριν και αν ε, δεν υπάρχει ανταπόκριση μπορεί κάποιος ε, να συμβουλευτεί τη βάση Eurodac, αλλά και πάλι προβλέπονται διάφοροι έλεγχοι στο σχέδιο, οι αρχές συντονισμού σε επίπεδο κράτος μέλος, οι αρχές επαλήθευσης που επαληθεύουν αν δικαιούται το κράτος μέλος να ζητήσει πρόσβαση και ούτω καθεξής. Υπάρχουν μέσα στο κείμενο πάρα πολλές τέτοιες ρήτρες. Ε, μιλάμε για πρόσβαση για τις αρχές επιβολής ε, νόμου, διότι είναι μια σύντομη έκφραση που μας βολεύει, αλλά ουσιαστικά ε, στέλνουμε ένα δακτυλικό αποτύπωμα απλώ ε, στην βάση Eurodac και περιμένουμε θετική αρνητική ανταπόκριση. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα στη βάση δεδομένων Eurodac και να ψάξει οποιοδήποτε δακτυλικό αποτύπωμα. Εσεί στέλνετε το δακτυλικό αποτύπωμα και βλέπετε αν υπάρχει μέσα στη βάση δεδομένων ή όχι. Ε, ξαναλέω ότι με χαροποιεί το ότι προβλέπεται και η Εθνική Βάση Δεδομένων και ε, η διαδικασία πριν εάν τώρα ένα κράτος μέλος δεν έχει ε, εφαρμόσει την ε, απόφαση πριν και θα ήθελα να ρωτήσω πόσα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει αυτή την απόφαση πριν μέχρι στιγμής και, ως, και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που εν μέρη έχουν εγκρίνει την απόφαση, δηλαδή στις σχέσεις τους με κάποια κράτη-μέλη και όχι με όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν τα κράτη-μέλη θα έχουν πρόσβαση στη βάση Eurodac. Στη συνέχεια ημερομηνίε. Ε, προτείνω τη 10η Οκτωβρίου για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσής μου, 18 Οκτωβρίου για την, ε, η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών. Ε, είναι προφανές ότι θα γίνουν συσκέψεις ανάμεσα στους Κιώδης και ψήφος ανατολισμού στις 27 Νοεμβρίου ενδεχομένως στην προβλεπόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Σας ευχαριστούμε κυρία Μακοβέλη Πρόεδρος. Σας ακούσουμε και άλλα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Γκίγιομ, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Μωράης που έπρεπε να τοποθετηθεί. Θα τα πω εγώ στη θέση του. Η Κομισιόν θύμισε την ε, μακρόχρονη διαδικασία για αυτό το κείμενο και τις περιπέτειές του τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θύμισε πολύ σωστά εξάλλου ότι αυτό το θέμα ε, θα έπρεπε να το εξετάσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πέρα δηλαδή από το άσυλο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις συλλογικά όλου του πακέτου άσυλο. Εγώ θα ήθελα τώρα να ρωτήσω μερικά πράγματα την Κομισιόν σχετικά με αυτό το θέμα. Το επίκεντρο της όλης προβληματικής είναι το θέμα της πρόσβασης της Ευρωπόλ στα, ε, στα φυσιές εσείς ε, αναφερθήκατε στο θέμα της διάσωσης αυτών των αρχείων. Θα θέλαμε όμως να ξέρουμε ποια είναι εκείνα τα ε, σημεία προστασίας, ε, τα σημεία που θέτουν όρια για την προστασία των δικαιωμάτων πρόσβασης στα αρχεία. Η διαχείριση των δεδομένων, η αξιοπιστία τους έχει αμφισβητηθεί αρκετές φορές από, πολιτι... από πολιτικά όργανα και εδώ ως Γαλλίδα εκφέρομαι Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα με την Eurodac για το θέμα της προστασίας των δεδομένων, έτσι το εξέφρασε δηλαδή ο Ευρωπαίος Ελεγκτής. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία για την Eurodac είναι πρόορη και υπάρχει ένας κίνδυνος άμα αρχίσουμε να συμμεριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες. Η πρόσβαση των δεδομένων στα δεδομένα, κυρίως αν αυτά είναι αναξιόπιστα, ε, πώς δίνονται εγγύησει. Με τις, όταν ζητώνται πληροφορίες ε, για τους ενδιαφερόμενους, πώς έχουμε εγγύησει ότι δεν ε, έχουμε επαφές και με τη χώρα προέλευσης και έχουμε δημιουργούμε ένα σύστημα καταστολής, μια δύναμη καταστολής. Διότι έχουμε από τη μια αυτούς ε, που ζητούν άσυλο και από την άλλη έχουμε το θέμα της εγκληματικότητας, το οποίο μπορεί να μαυρώνει αυτούς τους ετούντες άσυλο. Επίσης, αναφέρατε και, το θε... και την ε, τυπολογία παραδικήματος και θέλω να επανέλθω σε αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της, ε, του ευρωπαϊκού εντάλματος και θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Και έχω και πρόβλημα με μία φράση που λέει τα εξής η Ευρωπόλ μπορεί να συμβουλεύεται αυτά τα αρχεία για ειδικέ αναλύσεις ή ειδικέ αναλύσεις στρατηγικού τύπου. Για πέστε μου λοιπόν τι εννοεί αυτή η διατύπωση. Και ευχαριστώ κυρία Γκυγιόμ, η Λέδη Λότφορτ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι μαζί σας. Είχαμε ξανά προβλήματα με το ταβάνι του κτηρίου. του κτηρίου στο Στρασβούργο που έπεφτε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση αυτή μόνο και μόνο για να καλύψει τα κενά. Θέλω να πω ότι ικανοποιεί τα αιτήματα ορισμένων κρατών μελών και αποτελεί μέρος μιας διαπραγμάτευσης για τα μέτρα τα σχετικά με το άσυλο. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω τι προσφέρει σε αντάλλαγμα για αυτά τα μέτρα. Και αφετηρία μου είναι η θέση που πάντα είχα ότι με προβλημάτισε δηλαδή η πρόσβαση των αρχών επιβολής νόμου σε αυτά τα δεδομένα. Πιστεύω πως ε, αυτή η βάση δεδομένων είναι ξεχωριστή από ε, αυτήν εδώ την οποία συζητούμε. Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα αιτήματα για θεωρήσεις και αυτό με ανησυχεί. Με ανησυχεί. Με ανησυχεί λοιπόν η συνολική θεώρηση των ετούντων άσυλο ε, ως ε, πιθανούς εγκληματίες. Φυσικά, από την άλλη, υποστηρίζω την ανάγκη ασφαλιστικών δικλείδων και γι' αυτό καλωσορίζω τι γενικέ γραμμές της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί πιστεύω ότι έχουν εργαστεί αρκετά πάνω σε αυτέ τις ασφαλιστικές δικλίδες. Πραγματικά όμως να τονίσω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι η έσχατη λύση, όταν όλα τα υπόλοιπα μέσα που έχουμε στην έρευνα ενός εγκλήματος έχουν αποτύχει και φυσικά κρατώντας την αρχή του hit ή no hit, και την ανταλλαγή των δεδομένων αυτών με τις τρίτες χώρες. Κάτι που πιθανώς θα έθετε σε κίνδυνο τους ετούντες άσυλο. Το Συμβούλιο μπορεί να στηριχθεί στο Κοινοβούλιο στην υποστήριξη αυτών των ασφαλιστικών δικλείδων. Τώρα, δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το αν η συνθήκη του Προύμ είναι μία από τις προϋποθέσεις ή θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι το κείμενο, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να έχουν ψάξει προηγουμένως τις βάσεις δεδομένων των υπόλοιπων κράτων μελών σύμφωνα με τη συνθήκη Προύμ, όχι όλων των υπόλοιπων κρατών μελών. Και έχω εδώ τις ε, σημειώσεις των συζητήσεων του Συμβουλίου του Ιουλίου, όπου υπογραμμίζεται ότι τα κράτη, ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να Κοιτάξτε, εάν έχει γίνει έλεγχο σύμφωνα με την συνθήκη Προύμ και ακόμα και αν το κράτος μέλος αυτός δεν είναι συνδεδεμένο, δεν χρειάζεται να ψάξουμε σε άλλα, σε άλλες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών μελών. Όμως, ποιο είναι το εύρος της εφαρμογής της απόφασης αυτής σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια. Για μένα, η εφαρμογή του ΠΡΟΥΜ θα έπρεπε να είναι πλήρης. και όποιο κρατός μέλος επιθυμεί θα, μπορού, θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Eurodac. Χρειαζόμαστε πραγματικά να ελέγξουμε αυτό το σημείο. Επίσης, δεν με καθησυχάζουν τα σχόλια ορισμένων κρατών μελών στις συζητήσεις του Συμβουλίου όσον αφορά τις ε, ανάγκες για αυστηρές ασφαλιστικές ε, δικλείδες και την τήρησή τους για την αποφυγή περιπτώσεων παράνομης μετανάστευσης. Ναι, είναι πειρασμό. Όταν έχεις μια βάση δεδομένων μπορεί να έρθει κάποιος και να πει ας το κοιτάξουμε. Όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αναλογικότητα και η αναγκαιότητα. Και όσον αφορά την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα όσον αυτά για το πεδίο εφαρμογή. Τώρα όσον αφορά τις ε, εντεταλμένες αρχές. Στην απόφαση αυτή, ο κατάλογος των αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη-μέλη έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ίσως δεν ε, ή, δεν ξέρω, μπορεί να το έχω παραβλέψει εγώ, αλλά δεν βλέπω μια τέτοια διάταξη στην Eurodac Πιστεύω πιστεύω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Μετά, ορισμένα κράτη-μέλη συζητούν την ε, ιδέα να υπάρξει κάποια ετεταλμένη αρχή. Και εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να έχουμε ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης έτσι ώστε να ελέγχονται οι εκάστοτε αρχές επιβολής νόμου. Πιστεύω πως επίσης θα έχουμε συζητήσεις αν, όσον αφορά την πρόσβαση στην Ευρωπόλ και δεν μπορώ να καταλάβω εδώ που τα λέμε γιατί η Ευρωπόλ θα πρέπει να περνάει από εθνικό σημείο επαφής αντί να έχει πρόσβαση αμέσως το κεντρικό σημείο επαφής. Ίσως έχει να κάνει με την επαλήθευση των δεδομένων, όμως μου είναι ασαφές. Και θα είμαι σύντομη, διότι ο πρόεδρος θα με σταματήσει σε λίγο, αν συνεχίσω. Ε, ένα από τα σημεία που αναφέρθηκαν ήταν οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με το κανονισμό της Eurodac, να έχουν ήδη ελεγχθεί η βάση δεδομένων των ε, κρατών μελών σύμφωνα με το ΠΡΟΥΜ. Αυτό δεν προϋποθέτει πρόσβαση στην ΒΙΣ. Η, πρόσβαση, η απόφαση όμως ΒΙΣ είναι πρώτερη της απόφασης ΠΡΟΥΜ. Εν ολίγης αυτά για τις αρχικές μου απόψεις να τονίσω άλλη μια φορά ότι δεν με τρελαίνει αυτή η πρόταση. Φυσικά και εκτιμώ το σκεπτικό για την ανάγκη μιας τέτοιας ε, διαδικασίας για την ε, διερεύνηση εγκλημάτων. Αλλά βρίσκω ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική και πιο έντονη άποψη όσον αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες από κάποια άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τον κύριο Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και να πω και εγώ με τη σειρά μου πώς χαίρομαι που βρισκόμαστε πάλι εδώ και που θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές ήδη στο παρελθόν και θα ήθελα να αρχίσω με μια παρατήρηση που εμένα τουλάχιστον ε, με απασχολεί. Δηλαδή, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων, οι οποίες έχουν συσταθεί για έναν τελείω διαφορετικό σκοπό. Και η πρόσβαση αυτή στις αρχές επιβολής του νόμου δεν μου είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις αστυνομικές αρχές. Ποια πρότυπα ισχύουν. Και αυτό το λέω διότι ε, τώρα μόλις όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση Τη ε, προστασία προσωπικών δεδομένων που συζητείται στο Συμβούλιο και τη συνεργασία με τον αστυνομικό τομέα. Υπάρχει Υπάρχει, υπάρχουν, υπάρχει ένα μπλόκο, υπάρχουν εμπόδια στις ε, συζητήσεις αυτές και οδηγούμαστε σε πίσω γύρισμα. Αλλά πραγματικά πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, διασφαλίζοντας όμως την ε, τήρηση ορισμένων κοινών ελάχιστων προτύπων. Για την επαλήθευση των ετούντων άσυλο και την σωστή μεταχείρισή τους από τις αστυνομικές αρχές είναι φυσικά σημαντικό, όμως θεωρώ, το θεωρώ κάπως κοινικό και κάπως λάθος αυτή η πρόσβαση από τις αρχές να θεωρείται ότι γίνεται προς όφελος των ετούντων άσυλο είναι μια, η απόφαση του να χρησιμοποιούμε δεδομένα για διαφορετικούς ε, σκοπούς χωρίς να έχουν άμεση σχέση με τις αιτήσει ασύλου. Αυτό το θεωρώ... Θεωρώ μάλλον ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να καταστήσει σαφές ότι χρειάζεται μία ανάγκη για να γίνεται δυνατή η διαδικασία του hit ή no hit στις ε, αναζητήσεις αυτές. Επίσης, πρέπει να διατηρήσουμε τα κοινά ελάχιστα πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, την πρόσβαση σε δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Στο άρθρο της διατάξης, στο άρθρο 6 για, τις, ε, για τα verifying authorities. Αυτές οι αρχές επαλήθευσης, οι verifying authorities, για μένα ε, είναι οι δικαστικές, ε, για παράδειγμα, αρχές κατόπιν απόφασης δικαστηρίου. Εδώ αναφέρεται μια γενική υπηρεσία που θα είναι αρμόδια για, την, ε, για το να εξετάσει αν όλα αυτά συνάδουν με, τον κανονισμό. Αυτό όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί ποια θα είναι αυτή η αρχή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η πρόταση χρειάζεται ακόμα επεξεργασία. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Έχοντας ακούσει την κυρία Λάτφορντ, ε, ξέρετε, θα πω και εγώ ότι δεν πολύ ήθελα να έρθω εδώ πέρα, μήπως ε, πέσει το ταβάνι στο κεφάλι μας, ε, διότι ξέρετε ότι η δική μου η θέση είναι κάτω από εκεί που κατέβει το ταβάνι του κτηρίου του Στρασβούργου. Και... Ε, κάποιοι που θέλουν να υπερασπίσουν κάποια συμφέροντα και με σπρώχνουν να μπω σε άλλες θέσεις μου δημιουργούν ανησυχία και δεν πολύ ήθελα να έρθω εδώ. Μπα και συνέβαινε το ίδιο με αυτή την θέση. Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα πέρα από αυτό τις γενικές αρχές της ε, παρουσίασης ε, του νέου σχεδίου. Εγώ θεωρώ ότι ακούγονται λογικά αυτά για την προστασία των ετούντων άσυλο, αλλά ξέρετε με ανησυχεί αυτό που ακούγεται από κάποιου ότι παρόλε τι ρήτρε διαφύλαξης, εάν κάνουμε τη χρήση αυτών των ε, στοιχείων, εκμεταλλευόμαστε, και τονίζω αυτή τη λέξη, αυτούς που έχουν ζητήσει άσυλο. Εάν εξασφαλιστεί μια χρηστή διαχείριση, λένε κάποιοι, παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση αυτών των ετούντων άσυλο από εγκληματικά στοιχεία και άλλους που τώρα κάτι που τώρα συμβαίνει για και κάτι που θέλουμε φυσικά εμείς να καταστήλουμε. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ε, ακόμη και σε περιπτώσει όπου διευκρινίζεται για ποιο λόγο ένα κράτο ε, ζητάει στοιχεία. Όταν κοιτάζω τι κοινέ ερευνητικέ ομάδε, παραδείγματο χάρη, γιατί εγώ ήμουν αρμόδιο για αυτό το ζήτημα μέσω τη έκθεσή μου και διαπίστωσα πόσο δύσκολη ήταν η συνεργασία ανάμεσα στι αρχέ επιβολή νόμου. Αν όμω δεν εξασφαλιστεί η κατάλληλη συνεργασία με τι απαιτούμενε ε, δικλείδε ασφαλεία, υπάρχει σοβαρό κίνδυνο για καταχρήση. Ο κύριο Άλμπρεχτ το ανέφερε ανέφερε ακροφυγός. Πιστεύω ότι είναι καλό το σχέδιο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αυτές οι ρήτρε, αλλά δεν μας φτάνουν να μας ξεκαθαρίσει κάποιο ότι αφού θα τα έχουμε περάσει όλα αυτά, αφού θα, έχουν, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή ε, η περίπλοκη διαδικασία, θα γίνει επικοδομητική χρήση τη νέα ε, δυνατότητα από πλευρά των κρατών μελών για να ωφεληθούν αυτοί που αρχικά έπρεπε να ωφεληθούν με αυτή την πρόταση. Σα ευχαριστούμε κύριε Κύρκο, Ο κύριο Ντεγιούγκ τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ε, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την κυρία Γκυγιώμη και την κυρία Λάτφορντ για τον ε, ιονή στιγματισμό σε εισαγωγικά της ε, χρήσης της βάσης Eurodac. Αυτή ανέκαθεν ήταν η θέση της πολιτικής μας ομάδας διότι σε διάφορες χώρες και δυστυχώς και στη δική μου υπάρχουν πάρα πολλοί που σε καθημερινή βάση ε, απορρίπτουν ναι, τους ετούντες σε άσυλο και τους στιγματίζουν και, θα, και άρα ανέκαθεν να κατά μια τέτοια προσέγγισης. Τώρα, τίθεται ζήτημα ιδιωτική ε, ζωή και περιορισμού των ε, ατομικών ελευθεριών, οπότε θα πρέπει να αποδειχθεί ότι συντρέχει λόγο για να περιοριστούν αυτέ οι ελευθερίε. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους, δύσκολα μπορώ να φανταστώ εγώ μια κατάσταση όπου υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για την ε, ε, αρχή επιβολής νόμου για να έχει πρόσβαση στη βάση ε, δεδομένων. Έχετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα, υποθέτω. Όλοι έχουν όταν ερευνούν ένα έγκλημα. Έχει διαφύγει ο δράστης, ε, ας υποθέσουμε ότι έχει ζητήσει άσυλο σε κάποια άλλη χώρα, δεν ξέρω οι τρομοκράτες ή σοβαροί εγκληματίες για να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία του σχεδίου υπάρχουν. Εγώ, αν ήμουν τρομοκράτης ε, προσωπικά, ε, δεν θα δραπέτευα από ένα κράτος μέρος για να ζητήσω άσυλο από ένα άλλο. Είναι παράξενο και περίεργο και δύσκολο μπορώ να φανταστώ μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, στην αξιολόγηση αντικτύπου τη Επιτροπή δεν θα έπρεπε να μα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου θα υπάρχει αυτή η επιτακτική ανάγκη, θα συντρέχει ο λόγο για να γίνει χρήση τη νέα διάταξη. Επίση, ε, οι εντεταλμένε αρχέ, ποιε είναι αυτέ, προσοχή, είναι ε, εξαιρετικά γενικόλογη η διατύπωση προ το παρόν. Σα παραπέμπω επίση στο άρθρο 22 που έχει κέρια σημασία, διότι εκεί προβλέπονται οι όροι και οι προποθέσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Είναι εξαιρετικά κακή η διατύπωση. Έχουμε το εδάφιο 1α, όπου λέμε ότι <clears throat> για σκοπούς ε, έρευνας, ε, δίωξης ε, τρομοκρατικών εγκλημάτων, ενεργειών και συναφών εγκληματικών πράξεων, έτσι μας λέει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω όμως γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι πολύ γενικό λέει η διατύπωση. Και στο εδάφιο Β, ε, από νομική πλευρά, εφόσον είμαστε σε διαφορετικό εδάφιο, μιλάμε και για διαφορετικό, ε, είναι και διαφορετικό το αντικείμενο. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το δεύτερο εδάφιο και δεν έχω κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η νομική φρασιολογία. Ε, όπως είπα και στην αρχή, η πολιτική μου ομάδα ε, δεν μπορεί να εγκρίνει αυτή την πρόταση παρά μόνο αν περιοριστεί σε πολύ συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπρόνς. δεν μου συμβαίνει συχνά, αλλά συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη φορά. Ελπίζω να μην μου γίνει συνήθι. Λοιπόν, οι αρχές επιβολής νόμου μας λέει η Επιτροπή στα κράτη-μέλη που ερευνούν σοβαρές εγκληματικές ενέργειες θα έχουν πλέον το δικαίωμα να επαληθεύουν τα αποτυπώματα στην βάση δακτυλικών αποτυπωμάτων της Eurodac όπου έχουμε τα αποτυπώματα ε, των ετούντων ε, άσυλο. Λογικό μου ακούγεται αυτό. Επιβεβαιώθηκε δε, όπως ε, αν κατάλαβα καλά, ότι οι αρχές επιβολής νομού δεν θα μπορούν να μπαίνουν και να περιοδεύουν μέσα στην βάση δεδομένων ε, πρέπει πρώτα να έχουν στην κατοχή τους ένα δακτυλικό αποτύπωμα στο κράτος μέλος και στη συνέχεια να γίνει η επαλήθευση θετικής ή αντικής απάντησης. Hit ή no hit. Μόνο αυτή η δυνατότητα τους δίνεται. Είπανε κάποιοι ότι στιγματίζονται έτσι οι σε άσυλο. Όμως, εάν είχαμε βάσει δεδομένου με τα δακτυλικά αποτυπώματα των Ευρωβουλευτών, παραδείγματο χάρη. να μια καλή ιδέα για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιο αντίρρηση αν έχει ένα καλό λόγο ένα κράτο μέλο να ε, προσδοκεί μια θετική απάντηση, να έχει το δικαίωμα να κάνει την αναζήτηση δεν θα, ε, θα με εξέπλητε με μια τέτοια πρόταση, αλλά δεν θα με ενοχλούσε το να ελέγξει κάποιο ε, την βάση δεδομένων. Ο Γενικό Διευθυντή ε, τη Frontex νωρίτερα φέτο μα είπε ότι όσοι εισέρχονται παρανόμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφουν τα προσωπικά ταξιδιωτικά τους έγγραφα ε, προτού εισέλθουν στην Ένωση για να μην υπάρχει ε, κανένας ε, τρόπος να ξέρουμε από πού έρχονται. Λοιπόν, τα αποτυπώματα μας το επιτρέπουν. Γιατί όχι. Ωραία. Λέει ο Πρόεδρος, θα ακούσουμε την εισηγήτρια για, την, για τις παρατηρήσεις, αλλά έχουμε και τον Ευρωπαίο Επόπτη Δεδομένων εδώ, τον κύριο Χάστινγκς. Οπότε καλό θα ήταν ναι. Να τον ε, ακούσουμε... Να ακούσουμε ποια είναι η άποψή του. Πρωτού ακούσουμε και πάλι την εισηγήτρια. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία στις 5.30 και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό και εξάλλου έχουμε και άλλα ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε πριν τις 5.30. Ο κύριος Χάστινγκς, ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Την Τετάρτη μάλλον θα εκδώσω μια γνωμοδότηση με πολύ σημαντικά στοιχεία μέσα. Δεν θα είναι 100% θετική, να σας το πω αυτό. Αλλά θα σας δώσω τροφή για σκέψη. Θα δώσω σε αρκετές ομάδες τροφή για σκέψη. Πιστεύω όμως να δώσω προστιθέμενη αξία έτσι ώστε να βελτιωθεί αυτή εδώ η πρόταση. Και θα μιλήσω για το σύστημα ΑΣΥ στην επόμενη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάστινγκς. Κυρία Μακοβέ, επιστρέφουμε σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα όμως να ακούσω την απάντηση της Επιτροπής την ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπή. Ο κύριος Όιλ, αντιπρόσωπος της Επιτροπής, έχει σημειώσει τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία αναφερθήκατε. Πρώτου λοιπόν επιστρέψουμε στην κυρία Μακοβέη, θα παρακαλούσα να ακούσουμε τις απαντήσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις διατυπώθηκαν, θα προσπαθήσω να τις ε, καλύψω λακωνικά αλλά περιεκτικά. Καταρχάς, η κυρία Μακοβέη ρώτησε για την ε, συμφωνία Προύμ πόσα κρατημέλη την επικύρωσαν. Μέχρι τον Ιούνιο του 2012, 10 κρατημέλη την έχουν επικυρώσει στο πλαίσιο της χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και είμαστε αισιόδοξοι ότι τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες θα αυξηθεί ο αριθμός των κρατών μελών που θα την επικυρώσουν όσον αφορά την παρέμβαση του κυρίου Λάτφορντ. Έχετε δίκιο. Η επικύρωση πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να με να επικυρωθεί η συνθήκη Προύμ αλλά και να ε, δημιουργηθεί ένας, μια σύνδεση με, μόνο με κράτη-μέλη. Έπειτα, η κυρία Γκυγιόμ, έχει πολλές ερωτήσεις. Καταρχάς, όσον αφορά την πρόσβαση στην Ευρωπόλ, η πρόσβαση της Ευρωπόλ στην ε, βάση αυτή δεδομένων. Πιστεύουμε ότι δικαιολογείται το δικαίωμα πρόσβασης της Ευρωπόλ, διότι η Ευρωπόλ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος που αφορά ένα, ε, ε, δύο ή περισσότερα και συνδέει τις πληροφορίες που αντλεί από τα εκάστοτε κράτη-μέλη και τις αρχές επιβολής νόμου αυτών και με την διασταύρωση των πληροφοριών που λαμβάνει η Ευρωπόλη από τα διαφορετικά κράτη-μέλη θα μπορεί να έχει ξεκάθαρες ενδείξεις στην ε, αναγνώριση των ενόχων για διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Έπειτα, η κυρία Γκυγιόμ ρώτησε για τον ορισμό των σοβαρών εγκλημάτων και της τρομοκρατίας και πώς μπορούμε αυτό να το διατυπώσουμε σαφ... σαφώς. Στο άρθρο 2J γίνεται αναφορά στην τρομοκρατία και αναφέρεται η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου από το 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και όσον αφορά για τα σοβαρά εγκλήματα το άρθρο 2 παράγραφος K αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Υπάρχουν λοιπόν ξεκάθαρες αναφορές, συμπαγείς αναφορές σε ορισμούς σε αυτόν τον κανονισμό και σε αυτά τα σημεία. Κάτι άλλο τώρα που αναφέρθηκε όχι μόνο από την κυρία Γκυγιόμ αλλά και τον κύριο Άλμπρεχ και την Βαρόνη Λάμφορντ όσον αφορά τον στιγματισμό των ετούντων άσυλο. Πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να δούμε τα πράγματα με μια ευρύτερη προοπτική, να δούμε τις ασφαλιστικές δικλίδες που έχουμε εισαγάγει και να μιλήσουμε μόνο και το τονίσω αυτό, μόνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων όπως οι δολοφονίες. Υπάρχει κοινό συμφέρον να κλείσει αυτό το κενό που υπάρχει εδώ και εάν οι αρχές επιβολής νόμους αποκτήσουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση μόνο για αυτά τα σοβαρά ποινικά εγκλήματα, θα, μπορούν, θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους ενόχους. Και πιστεύω ότι θα, αυξηθεί, θα αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχία τους. Δεν θα στιγματιστούν οι ετούντες άσυλο, διότι σε πρώτο στάδιο υπάρχει μόνο ένα δακτυλικό αποτύπωμα, το οποίο βρέθηκε σε μια σκηνή εγκλήματος και το οποίο θα στέλνεται στην Eurodac. Δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα παραπάνω, δεν υπάρχει όνομα, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον ετών άσυλο. Μόνο εάν υπάρχει θετική απάντηση, μόνο εάν υπάρχει hit σε αυτό το δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε σε μία σκηνή ε, σοβαρού εγκλήματος. Μόνο λοιπόν τότε, εάν αυτό το δακτυλικό αποτύπωμα ε, έχει θετική ανταπόκριση από την βάση Eurobac, τότε θα υπάρχει συνέχεια τότε θα ζητηθούν ενδεχομένως λεπτομέρειες και ενδεχομένως υπάρξει ανταλλαγή περαιτέρω δεδομένων. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν αντιπαραθέσουμε το συμφέρον για την, ε, για επίλυση και την ε, διερεύνηση των ε, σοβαρών εγκλημάτων και αυτή την πρόταση, θα δούμε ότι υπάρχει μια ισορροπία και την πρόταση είναι ισορροπημένη. Έπειτα. Βαρόνι Λάτφορντ, νομίζω ότι απάντησα τις περισσότερες ερωτήσεις σας. Ε, είπατε ότι πρέπει να είναι έσχατη λύση ασφαλιστικές δικλείδες και αυτό είναι ουσιώδες σημείο στην πρότασή μας. Έπειτα, οι αρχές που θα οριστούν, θα δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα. Εδώ να σας παραπέμψω στο άρθρο 40 ή 4 όπου αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ειδοποιούν τις εντεταλμένες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δημοσιευθεί αυτό στην επίσημη κοινοτική εφημερίδα. Πρόεδρος, κύριε Όλη, σας παρακαλώ να συντομεύετε γιατί πρέπει να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Δύο σημεία έχουμε να συζητήσουμε πριν την ψηφοφορία. Νομίζω πως τελείωσα. Σχεδόν. Όσον αφορά την ε, σύνταξη του άρθρου 20, η κυρία Κιγιόμ ανέφερε ότι όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να αναφέρονται στο άρθρο 20. Πρέπει να πληρούνται λοιπόν όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Και αυτά προς το παρόν. Να ζητήσω συγγνώμη αν ξέχασα κάτι. Κυρία Μακοβέη, πίσω σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πως πρέπει να είμαι σύντομη. Θα συζητήσω με τους συναδέλφους μου για τις ανησυχίες τους, για τις ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά πιστεύω ότι η Επιτροπή πραγματικά θα ε, λάβει υπόψη τις ασφαλιστικές δικλίδες που πρέπει να υπάρχουν. Όμως, αν οι συναδελφοί μου έχουν κάποια περαιτέρω σχόλια, με τα χαράς να τα συζητήσω μαζί τους. Τώρα, όσον αφορά την έσχατη λύση, ναι, έσχατη λύση. Θα κοιτάξουμε πρώτα τι εθνικέ βάσει δεδομένων και μετά τι υπόλοιπε. Και αν υπάρχει θετική απάντηση, αν υπάρχει χ, τότε μετά θα ρωτήσουμε, οι αρχέ μάλλον επιβολή νόμου, θα ε, ζητήσουν ε, απάντηση από την βάση Eurodac. Συνάδελφε, μας δώσατε ένα παράδειγμα και θα ήθελα να σας δώσω εγώ με τη σειρά μου ένα παράδειγμα χρήσης. Για παράδειγμα, σκηνή εγκλήματος διαπράτεται ένα σοβαρό έγκλημα. που υπάγεται στα πλαίσια της οδηγίας για την τρομοκρατία. Σε αυτή τη σκηνή λοιπόν του εγκλήματος συλλέγονται τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τα, κοιτά, τα ψάχνετε στην δική σας Εθνική Τράπεζα Δεδομένων, ψάχνετε και σε άλλες και μετά χρησιμοποιείτε την ε, Συμφωνία Προύμ και εάν δεν βρείτε κάτι τότε ζητάτε από την Eurodac απάντηση. Τότε στέλνετε το αποτύπωμά σας στη Eurodac και ζητάτε θετική ή αρνητική απάντηση. Και μετά, εάν υπάρχει θετική απάντηση, τότε παίρνετε ε, το όνομα μιας χώρας και χρησιμοποιείται η αρνητικη απαντηση και μετα εαν υπαρχει θετικη απαντηση τοτε παιρνετε το ονομα μιας χωρας και χρησιμοποιειτε η αρχη της ε, αμοιβαία ε, εξυπηρέτησης. Ζητάτε λοιπόν από την Eurodac να σας πει σε ποια χώρα πρέπει να απευθυνθείτε. Δεν ζητάτε απάντηση από 27 διαφορετικά κρατημέλη που είναι αυτό που γίνεται τώρα. Θα πλουστευτεί η διαδικασία για αυτό το δακτυλικό αποτύπωμα. Ξανά λοιπόν όσον αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες, καλωσορίζω τις προτάσεις των συναδέλφων εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αρκούν αυτά. Έχουμε πρόσφορο έδαφος για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας περάσουμε και στο επόμενο σημείο για να προλάβουμε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμμετοχή σας, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση και τώρα θα περάσουμε ε, στα σημεία που σχετίζονται με το Σέγγεν. Το σημείο 6 πρώτα απ' όλα σχετικά με την ε, μετάβαση από το σύστημα ε, ΣΥΣ SIS-1 στο σύστημα πληροφοριών ε, του Schengen δεύτερης γενιάς, δηλαδή SIS-2, αναδιατύπωση. Ο κύριος Κάλλος Κοέλιο είναι ο εισηγητής μας. Θα μας κάνει μια γενική επισκόπηση και στη συνέχεια θα ακούσουμε την παρουσίαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα επόμενα πέντε λεπτά σα παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι στι 5.30 θα ψηφίσουμε και προτείνω μετά την παρέμβαση του εκπροσώπου ή τη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσουμε και τον κύριο Χάστινγκ, στον Ευρωπαίο Επόπτη και Μετά την παρέμβαση του κυρίου Κοέλιο θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα η Επιτροπή θα κάνει την παρουσίαση από ό,τι κατάλαβα. Ο κύριος Τιούντεραχ εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, λιγότερα από πέντε λεπτά μάλιστα. Περί τίνος πρόκειται. Ο στόχος της αναθεώρησης είναι σαφής. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να εγχύσουμε νομική ασφάλεια και προβληψιμότητα στα, ε, ως προς τη μετάβαση. Γιατί τώρα και όχι το 2008 όταν εγκρίθηκε το πρώτο νομοθέτημα για τη μετάβαση στο νέο ε, σύστημα. Αυτό έγινε διότι δεν είχαν ξεκαθαριστεί τα πράγματα, ε, το οποίο και συνέβη από το 2008 μέχρι το 2011. Διευκρινίστηκε λοιπόν η τεχνική διαδικασία ε, με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και μόλις ολοκληρώθηκε, δηλαδή μόλις ε, διευκρινίστηκε και με ποιο τρόπο όλα τα κράτη-μέλη θα μεταβούν στο ΣΥΣ 2, προέκυψε με σαφήνιο ότι χρειάζεται προσθήκη νομικής ασφάλειας στην όλη διαδικασία και τα κράτη-μέλη που θα ε, μετέβαιναν πρώτα στο νέο σύστημα χρειάζονται φυσικά νομική βάση Παρκώ ξεκάθαρη. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Τιούντεραχ, ένα λεπτάκι. Ε, υπάρχουν κάποιοι που έκαναν ένα πηγαδάκι στο μέσο του διαδρόμου και δεν υπάρχει ησυχία. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να ακούσουμε τον κύριο Τούντεραχ. Συνεχίζουμε. Ε, Χρειάζεται και να προσθέσουμε αυτό το στοιχείο της νομικής ασφάλειας στην ε, τεχνική διαδικασία και πιστεύουμε ότι με την ε, νέα διατύπωση τα καταφέραμε. Επίσης φαίνεται ότι τώρα σε τεχνικό και σε νομικό επίπεδο συμφωνούμε και με τα κράτη-μέλη ότι έχει επιτευχθεί αυτό. Δεύτερος στόχος αυτής της πρότασης ήταν να προσθεθεί η δυνατότητα εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας για κάποιες εθνικές δραστηριότητες μετάβασης προς το σύστημα Νέα γενιά, όπως η χρήση του EBF παραδείγματο χάρη, ακόμη και αν ναι, γίνει ε, αυτό αν αφορά αυτό στο τέταρτο σημείο, κάτι που συνέβη προ τη έγκριση του νέου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που ε, θέλουν να μεταβούν στο σύστημα ΣΥΣ2 και ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτή είναι η τελευταία φάση προτού τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα και άρα θα καθυστερήσει η όλη διαδικασία διότι δεν υπάρχουν πόροι για κάποια κράτη-μέλη για να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες της μετάβασης προβλέφθηκε αυτή η οικονομική βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω και μια σύντομη παρουσίαση για το ΣΥΣΕ2, διότι έχει ιδιαίτερη σημασία κατ' εμέ ε, σε αυτό το πλαίσιο να γνωρίζουμε. Πρώτον, ότι έχουμε εισέλθει στο τελικό στάδιο δοκιμών του ΣΥΣΕ2. Γνωρίζω ότι ε, τα τελευταία χρόνια ακούγονται πολλά για τις δοκιμές ε, του ΣΥΣΕ2. Το Μάιο το Master 2 ε, με επιτυχία. Αυτή είναι μία από τις προϋποθέσεις που έθεσαν τα ίδια τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου για να συνεχιστούν συνεχιστεί η τεχνική ε, διαμόρφωση του προγράμματος ως είχε, ε, θα, περισσότερες λεπτομέρειες ε, θα έχετε στην εξάμενη έκθεση που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά θα κοινοποιηθεί και στο Κοινοβούλιο. Έχουμε και τις συνολικές δοκιμές. Έχουμε το, την τελευταία σειρά δοκιμών ε, που θα ολοκληρώσει το σύνολο των δοκιμών ε, για το σύστημα 2 και θα εισέλθουμε στην ε, τελευταία πραγματική φάση που είναι η μετάβαση, η ίδια η μετάβαση στο ΣΥΣ 2. Εξού και ο επίγον χαρακτήρας του ζητήματος θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν, ε, διότι χρειαζόμαστε τη νομική βάση που υπάρχει μέσα στη νέα πρόταση, ούτω ώστε να ολοκληρώσουμε την φάση μετάβαση. Σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Χάστινγκ ε, τώρα ε, θα μα δώσει την άποψή του για αυτό το ζήτημα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα υπάρξουν πολλές περιστάσεις του επόμενου μήνε όπου θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα τη προστασία των δεδομένων. Τώρα εξετάζουμε μια ειδική διάσταση. Μιλήσαμε για το Eurodac, αλλά τώρα μιλάμε για ένα άλλο παράδειγμα. Πρόκειται λοιπόν για τη μετάβαση στο SIS2. Είναι μια διαδικασία κέρια σημασία. Είναι εξαιρετικά περίπλοκη αυτή η τεχνική διαδικασία και ενέχει και κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου. Ε, επί τη βάση της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι την καλωσορίζω διότι επιφέρει βελτιώσεις. Καλωσορίζω όλους ιδιαίτερο συγκεκριμένο ότι διευκρινίζει την εφαρμοσιμότητα του κανονισμού ΣΥΣ 2 ε, από την πρώτη μετάβαση από πλευρά κράτους μέλους και μετά. Αλλά ας περάσουμε τώρα στους ειδικούς ε, κινδύνους που ενέχει η διαδικασία. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μας πέντε περίπου ζητήματα που δεν έχουν ε, ε, διευκρινιστεί επαρκώς και αυτό ε, αιτιολογεί και μία γνωμοδότηση που εξέδωσα τον Ιούλιο και την οποία απλώς θα συνοψίσω εδώ. Το πρώτο σημείο είναι το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού μετάβαση. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο, απολύτως ξεκάθαρο το πεδίο. Κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιες κατηγορίες θα κάνουν την μετάβαση και ποιες όχι. Εάν ε, επίσης η μετάβαση ε, συνδέεται με, με τα ποιήση στοιχείων, ε, δηλαδή φόρτωμα δεδομένων και μεταφορά του από το ΣΥΣ1 και ΣΥΣ2 και τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα δεδομένα που δεν θα μεταναστεύσουν, δεν θα μεταφερθούν σε, σε αυτό το νέο σύστημα. γιατί συμβαίνει με τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί αλλά παρόλα αυτά παραμένουν μέσα ε, στον εξοπλισμό του ΣΥΣΕΝΑ. Είναι κάποια τεχνικά ζητήματα τέτοια φύσεω ε, που θα πρέπει να διευκρινίσουν. Έχουμε του ε, μηχανισμού ανάθεση ε, από την κοινή εποπτική αρχή. Πρέπει να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ακριβώ επειδή είναι εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία και άρα θα συμβουλεύαμε το εξή εξ αρχής, από την αρχή της διαδικασίας, ε, να εκινήσει και αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Σας ενημερώνω ότι σκοπεύουμε να κάνουμε μια, ένα ολοκληρωμένο έλεγχο ασφάλειας της κεντρικής ε, μονάδας, ε, καθώς και των προγραμμάτων μελλοντική εξέλιξη, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ΣΥΣ2 για όλα τα επόμενα στάδια. Τρίτον, οι διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων πρέπει να καταγράφονται κατά το δέον. Στο άρθρο 15 επαναλαμβάνει αυτό το σημείο, δηλαδή ότι οι ε, συνήθεις διαδικασίες οφείλουν να καταγράφονται. Όμως εδώ ε, μιλούμε για τη διαδικασία μετάβασης η οποία έχει κινδύνους, άρα και εκείνη πρέπει να καταγραφεί. Σημείο 4. Ο ρόλος και τα, τα κριτήρια αξιολόγησης ε, για να διαπιστώσουμε αν ήταν επιτυχής μετάβαση ή όχι. Στην ανάλυση μας είδαμε κάποια ασαφή ε, ζητήματα, ασαφή ως προς ε, την σαφήνεια που μπορεί να προσδοκά κανείς από μία αξιολόγηση. Νομίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τα κριτήρια ε, αξιολόγησης. Γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο που δεν επιτυγχάνει η μετάβαση. Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο Β. Δεν θα πρέπει όμως να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν είναι σαφές ποια διάταξη είναι εφαρμόστη. Κατόπιν, οι βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε ε, στις τεχνικές διατάξεις. Η απέτηση για την διεξαγωγή αξιολόγηση ε, κινδύνου και κατάρτιση σε σχεδίο αντιμετώπιση του εντοπιστέντο κινδύνου είναι δύο στοιχεία απαραίτητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβέστερα την πολιτική ασφαλείας για το σύστημα ΣΥΣ2 προτού αρχίσει η μετάβαση και όχι να γίνει πρώτη μετάβαση και μετά βλέπουμε. Μέσα στην γνωμοδότησή μου πραγματεύομαι διεξοδικά ε, αυτά τα επιμέρους ζητήματα. Τώρα θα μπορούσα να πω συνοπτικά ότι στο όλο εγχείρημα δεν μπορούμε να αφήνουμε στην τύχη κάποια πράγματα και ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιμείνει και για τα δύο. Και ε, να διευκρινιστεί η διατύπωση του κειμένου και να προσδιοριστούν λοιπά μέτρα που θα καλύψουν τους περιορισμούς του αναθεωρημένου ε, σχεδίου κανονισμού. Αυτά τα δύο ζητήματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα. Σας ευχαριστούμε κύριε Χάστινγκς, λέει ο Πρόεδρος. Ακούσαμε την γνωμοδότηση του επόπτη προστασίας δεδομένων. Δεν ξέρω τώρα, άλλαξε ο εκπρόσωπος Πρωτό ακούσουμε τον εισηγητή μας. Θέλετε από πλευράς του Συμβουλίου μήπως να παρέμβετε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η πρόταση για τη μετάβαση από το σύστημα συς 1 στην δεύτερη γενιά γενιά 2 παρουσιάστηκε στα κρατημέλη τον Μάιο του 2012 και από τότε το Συμβούλιο, κάτω από την Κυπριακή Προεδρία, εργάστηκε με τα κρατη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σταθεροποιήσει και να ενοποιήσει το κείμενο και τις προτάσεις έτσι ώστε καταρχάς να λάβει υπόψη τις θέσεις των ε, κρατών μελών και να αντικατοπτρίσει την ε, συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στο σύστημα αυτό και να εγγυηθεί την ε, ακρίβεια στις ε, τεχνικές ε, προδιαγραφές ορίζοντας τις επιμέρους ε, τεχνικές ομάδες επιγνώμενων από το εκάστοτε κράτος μέλος. Η πρόταση αυτή συζητήθηκε σε διάφορα επίπεδα στο Συμβούλιο. κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία για το κείμενο, το οποίο τώρα είναι έτοιμο προ υιοθέτηση. Η Κυπριακή Προεδρία γνωρίζει την σημασία, τη μεγάλη σημασία του νομικού αυτού οργάνου για την περάτωση του συστήματος ΣΥΣ2 και έχει εργαστεί για την ολοκλήρωση του φακέλου αυτού σε επίπεδο Συμβουλίου. Είναι ε, κατόπιν αυτού ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ε, διαβούλευσης. Αναμένουμε την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Κοέγιο, η σειρά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχίζοντας να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίαση της ε, πρότασης, να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Πίτερ σε τον Ευρωπαίο Επόπτη Δεδομένων, για την γνωμοδότηση που εξέδωσε για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να συγχαρώ φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Από ό,τι φαίνεται τελικά θα αποκτήσουμε ένα σύστημα πληροφοριών νέας γενιάς, δεύτερης γενιάς ε, του Σέγγεν. Ε, Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο ε, πολύ σημαντικέ δοκιμέ και έχω την εντύπωση ότι μπορεί να αρχίσει ε, το σύστημα να λειτουργεί από τον Ιανουάριο και το ΣΥΣ2 να λειτουργεί πλήρω από τον Απρίλιο του 2013 και μετά. Πολύ καλά νέα, πολύ καλά νέα για όλου όσου ε, συμμετείχαν στην συνολική προσπάθεια και αυτό που μας ικανοποιεί όλου ιδιαίτερω είναι πρώτον ε, ενισχύεται η ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την χρήση του νέου συστήματος. Δεύτερον, ε, η προστασία δεδομένων ανέρχεται σε ένα νέο υψηλότερο επίπεδο και τρίτον, αυτά που ε, αποτελούσαν αντικείμενο διαχείριση σε διακυβερνητικό επίπεδο πλέον ε, περνάνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο χάρη σε νέα τεχνολογικά εργαλεία που δημιουργούμε, όπως εξάλλου ήθελε ανέκαθεν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν γέννη διακύμεθα θετικά υπέρ της ε, πρότασης αυτής, όπως και υπέρ όλων των νομοθετημάτων που ρυθμίζουν αυτή τη μετάβαση από το ΣΥΣ1 στο ΣΥΣ2 και όπως τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ο κύριος Χάστινγκς μας ικανοποιεί το ότι η πρόταση για, το νομικό, για την νομική βάση του ΣΥΣΕ 2 θα έχει άμεση ισχύ στο πρώτο κράτος μέλος που θα κάνει την μετάβαση προς το ΣΥΣ 2. Αυτό μας εξασφαλίζει ε, ενισχυμένη ε, νομική ασφάλεια, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, το επίσης πάρα πολύ θετικό είναι θα βοηθηθούν οικονομικά τα κράτη-μέλη για να περατώσουν την μετάβαση στο ΣΥΣ 2. Εάν λοιπόν ε, κάποιο κράτος μέλος δεν διαθέτει τους πόρους και για να κάνει σε την μετάβαση προβλέπεται πλέον οικονομική βοήθεια, κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Ε, βλέπουμε ότι δεν έχουμε χρόνο συνήθως. Ε, ζητώ τη συνεργασία των συναδέλφων ε, ούτω ώστε να προχωρήσουμε για να είναι έτοιμο το νομικό πλαίσιο και τα κράτη-μέλη που είναι έτοιμα και το επιθυμούν να έχουν εγκαίρω στη διάθεσή του τα απαιτούμενα κονδύλια και το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσουν το νέο σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάλι θα ε, αποδείξει ότι δύναται με ταχύς ρυθμούς να προβαίνει σε αποφάσεις και δεν θα μπορέσει ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο να μας καταλογίσει η ολιγορία, η καθυστέρηση σε σχέση με μια πρόταση που προωθούν. Ε, τώρα, ε, λυπούμε, για να περάσω στα αρνητικά, ε, για το ότι μια τέτοια πρόταση με τόσο μεγάλη δημοσιονομική επίπτωση δεν έχει μια, δεν υπάγεται σε μια ενίσχυση, σε μια συγγνώμη ενισχυμένη διαδικασία διαβούλευση. Ε, τώρα, σε σχέση με την ημερομηνία θέσης ε, σε εφαρμογή, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη και από ό,τι ακούω είναι ότι θα είναι λοιπόν λειτουργικά τα εθνικά συστήματα τον Απρίλιο του 2013, δεν βλέπω καμία δυσκολία να προβλέψουμε ε, ως ημερομηνία τον Ιούνιο του 2012 είναι ένα από τα ζητήματα που συζητούμε με τους σκιώδεις εισηγητές μας, αλλά πάντως για την σκοπούς ε, προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων και των ατομικών ε, δικαιωμάτων ε, όπως μας είπε και ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, κύριος Χάστινγκς, οφείλουμε όλοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας ώστε να ολοκληρωθεί ε, το εγχείρημα. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο και τώρα θα συνεχίσουμε με τα μέλη της Επιτροπής που επιθυμούν να παρέμβουν. Η Βαρόνι Λάτφόρτ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση προς επιβεβαίωση. Η Προεδρία ανέφερε και από ό,τι καταλαβαίνω το Συμβούλιο, η νομική μάλλον υπηρεσία του Συμβουλίου, μετά από συνεργασία με την Επιτροπή και ελπίζω, κύριε Κόλλιο, να μου πείτε και εσείς ότι είστε ευχαριστημένος με αυτό. Το Συμβούλιο, λοιπόν, οι νομικές υπηρεσίες έχουν συμφωνήσει να χωρίσουν την πρόταση στα δύο. Το ένα μέρος να ασχολείται με το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλλον και η Ιρλανδία συμμετέχει, θα δεν μπορεί μάλλον να συμμετέχει ως ε, μη μέλος του Σέγγεν. Μπορείτε λοιπόν να μας επιβεβαιώσετε ότι αυτό ισχύει. Πιστεύω πως σε γενικές γραμμές αναφερθήκατε σε ορισμένα μέτρα, σε ορισμένες διατάξεις που θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ιρλανδία. Δεν ε, Μας αναφέρατε όμως τι θα γίνει, αν πραγματικά θα διαχωριστεί αυτό το νομικό όργανο. Δυστυχώς, καμία κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τώρα δεν έχει συμφωνήσει με τις απόψεις μου στο θέμα αυτό του Σέγγεν. Αυτά, κύριε Λάτφορντ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κοέλιο επίσης. Η πράσινη με σκιώδη συγκητή τον κύριο Νόκα, ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εμείς λοιπόν ως πράσινοι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την θέση σας. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη τα ζητήματα τα οποία έθιξε και ο κύριος Χάστινγκς είναι ιδιαίτερη ε, ζωτική σημασίας και ελπίζουμε επιτέλους αυτό το έπος να λάβει ένα τέλος. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Κέλλερ. Κύριε Λάτφορντ, διατυπώσατε ένα ερώτημα στην Κυπριακή Προεδρία. Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως είναι καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τις εξηγήσεις σχετικά με αυτόν τον διαχωρισμό των εγγράφων. Μάλιστα, η Επιτροπή έχει το λόγο τότε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν... Θέλω να πετάξω τον παλάκι, αλλά δεν ήμασταν εμείς που προτείναμε το διαχωρισμό, όμως ναι, υπάρχει ένας διαχωρισμός. Ευχαριστώ. Γκίγιομ, θέλετε το λόγο. Λυπούμε, εγώ σήμερα είμαι το τσιράκι των συναδέλφων. Αυτή την εντύπωση έχω, αλλά ο συνάδελφος ήθελε να μιλήσω εγώ στη θέση του και ήθελε να, έχει, να ξέρει τι γίνεται, ποιο είναι το καθεστώς της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, γιατί δεν διευκρινίζεται αυτό μέσα στη θέση. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Επιτροπή δεν θέλει να απαντήσει στην ερώτηση για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Θα κάνω τα τελικά σχόλια, λοιπόν, αν συμφωνείτε. Επιτροπή πάλι. Μάλιστα, φυσικά το ζήτημα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας πρέπει να ξεκαθαριστεί όσον αφορά την ένταξη στο σύστημα. Όλες οι χώρες θα αντιμετωπίζονται όπως, όλοι, όπως ήθιστε. Φυσικά πολιτικά έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν σε αυτό το σύστημα. Έχουν γίνει τεστ, έχουν εξεταστεί. Η τελευταία περίοδος ε, που διεξάγονται τα τεστ γίνεται τώρα και μετά θα είναι έτοιμα αυτά τα κράτη όταν πολιτικά το θελήσουν να ενταχθούν στο Σέγγεν 2. Κύριε Κοέλιο, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω μόνο αυτά που υπόθηκαν σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει στο ΣΥΣ2. Θα έχει βέβαια πρόσβαση μόνο στους ε, συναγερμούς. Όσον αφορά τις προτάσεις, θα στείλω στους σκιώδεις εισηγητές αυτή την εβδομάδα τις τροπολογίες μου για να επιτευχθεί μια συνένεση ανάμεσα στους κοιόδης εισηγητές και να ληφθούν υπόψη τα μεγαλύτερα ε, κομμάτια των ε, προτάσεων που έγιναν έτσι ώστε να τα βάλουμε στην ημερήσια διάταξη την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτά λοιπόν προς το παρόν για αυτό το θέμα. Τώρα μπορούμε να θέσουμε τις προθεσμίες για τις τροπολογίες για την επόμενη συνεδρίαση λοιπόν της Επιτροπής μας, της ΛΥΜΠΕ, τον Σεπτέμβριο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου και τότε θα παρουσιαστεί και το σχέδιο έκθεσης. Προχωράμε. Ίσα που προλαβαίνουμε στο επόμενο σημείο μέχρι να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία που προβλέπεται για τις 5.30. Το σημείο 7. Η θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων, το Eurosur. Εισηγητής κύριος Μάλντερ, Γιάνν Μούλτερ. Και εδώ, σε αυτή την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, θα έχει τη δυνατότητα η Κυπριακή Προεδρία και η Επιτροπή να τη σχολιάσει και φυσικά τα αγαπητά μέλη να λάβουν το λόγο. Κύριε Μούλτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα τοποθετήθηκα σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της αρχής. Ε, είμαι υπέρ σε μεγάλο βαθμό. Εάν έχετε ένα ευρωπαϊκό χώρο που μπορούν να μετακινηθούν οι πολίτες, είναι απαραίτητο να προστατεύεται και τα εξωτερικά σύνορα. Η πρόταση για το Eurosur που θα είναι τμήμα της Frontex θα έχουμε έναν εθνικό κέντρο συντονισμού και το κεντρικό συντονισμό σε επίπεδο Frontex. Νομίζω ότι όλες αυτές οι ιδέες μπορούν να τύχουν της υποστήριξής μας, όμως έχω και σοβαρές ανησυχίες. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι από τα πράγματα που με ανησυχούν περισσότερο από όλα. Ε, οι άνθρωποι μετα... Ε, ταξιδεύουν και πεθαίνουν σε μικρές βάρκες, σε μικρά φουσκωτά και κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται. Τέτοιες τραγωδίες πρέπει να τις αποφύγουμε και ε, γι' αυτό το λόγο προτείνω να καταστεί αποτελεσματικότερο το Eurosur. Πρώτα απ' όλα δεν επαρκεί να εξετάζουμε την κατάσταση αποκλειστικά και μόνο στα δικά μας εξωτερικά σύνορα. Πρέπει ταυτόχρονα να συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε χώρες όπου οι εξελίξεις ε, μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση που επικρατεί στα δικά μας εξωτερικά σύνορα. Στις ε, περισσότερες χώρες του κόσμου έχουμε αντιπροσωπεία, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δηλαδή εκπροσωπείται. Εγώ προτείνω να ενισχυθεί την περαιτέρω συνεργασία με τις επιτόπου αντιπροσωπείες και όχι μόνο να λαμβάνουμε πληροφορίες από τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού αλλά και από ε, κάποια ε, στελέχη της αντιπροσωπείας ε, της εξωτερικής δράσης ε, στην Αλγερία, στην Τινησία, στην Ουκρανία, οπουδήποτε. Δεύτερον, προτείνω στενότερη συνεργασία με εφιστάμενους οργανισμούς, παραδείγματο χάρη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ή Ελέγχου της Αλίας. Έχετε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δορυφορικών Στοιχείων που εδράζεται ε, στην ε, Μαδρίτη και οι τρεις αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τους μετανάστες και πληροφορίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την προστασία των εξωτερικών μας ε, συνόρων. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλλει στην ενημέρωσή μας και στην ε, μελλοντική δράση του Frontex. Άρα προτείνω καλύτερη χρήση των ε, υποδομών που διαθέτουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχουμε καλύτερη ενημέρωση ως προς την κατάσταση που επικρατεί στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Επίσης, πρότεινα και απευθύνω έτσι ένα αίτημα προς τα κράτη-μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία να μπορέσουν να συμμετάσχουν παρότι δεν ε, ανήκουν στο Σέγγεν, διότι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να μετάσχουν στο σύστημα Eurosur και θα έπρεπε να το καλωσορίσουμε αυτό το αίτημά τους. Ισχύουν τα συνήθη εχέγγυα φυσικά, αλλά χρειαζόμαστε ίσως περισσότερη προσοχή για τις ε, καταχρήσεις. Να τα θέσουμε μια τροπολογία, παραδείγματος χάρη, που να λέει ότι ε, τέτοιε πληροφορίε που έχουν συλλεχθεί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαβαστούν σε τρίτε χώρε, θα παραμείνουν ε, στι υπηρεσίε πληροφοριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η ενημέρωση, οι πληροφορίε, οι όποιε πληροφορίε ε, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα εξωτερικά σύνορα. Αλλά ε, ξέρετε, έχουμε πολλά σημεία εξόδου. Έχουμε τι αερολιμένε, έχουμε τα σημεία διέλευση των χερσαίων σύνορων. Δεν πιστεύω ότι ενδείκνεται τώρα ο χρόνο να συμπεριλάβουμε ε, νέα διάταξη γι' αυτό, αλλά αν κάποια κράτη-μέλη θέλουν να κινηθούν ταχύτερα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδιστούν λόγω ε, της ε, νέας ε, πρότασης. Αυτά θα ήθελα, ε, Πρόεδρε, να σχολιάσω προς το παρόν ως προς την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κύριο Όλιβερ ε, Σάιφελτ. Ευχαριστώ. Ε, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο έκθεσης για τη σαφήνεια και το όρομα που προσφέρει ως προς την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Θα ήθελα να δώσω τρία σύντομα παραδείγματα που είναι όμως παραστατικά. Πρώτον, προστασία των μεταναστών. Πρέπει στη, κατά την ε, προστασία των εξωτερικών μας συνών αυτό να αναδειχθεί σε προτεραιότητα και όχι να επικεντρωνόμαστε ε, σε, στα προληπτικά μέτρα, δηλαδή την αποτροπή του διασυνοριακού εγκλήματος ε, και την παράνομη είσοδο κάποιων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή, αυτή πρέπει να είναι η πραγματική στόχη του Eurosur. Ο κύριος Μούλτερ ανέφερθηκε στα, φουσκωτά, τα μικρά σκάφη με τα οποία μεταφέρονται οι λαθρομετανάστες. Ε, αυτό το σημείο το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν αυτά τα μικρά σκάφη αλλά αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτος ο απολογισμός νεκρών, κυρίως στη Μεσόγειο, όπως ανέφερε ο κ. Μούλτερ. Δεύτερον, έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια στο νέο άρθρο 12α για την προστασία των δεδομένων χάρη στην πρόταση του κυρίου Μούλτερ. Διευκρινίζεται σε ποιε περιπτώσει μπορούν ε, να ανταλλαχθούν τέτοια στοιχεία υπό ε, ε, αυστηρού νομικού περιορισμού. Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων δεν είναι στόχο του Eurosur, αλλά όπω έλεγα. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση του κ. Μούλτερ προσδιορίζει ποιε πρέπει να είναι αυτέ οι εξαιρέσει στο γενικότερο κανόνα. Τρίτον, το σχέδιο έκθεση έχει σαφέστατο όραμα σε σχέση με το Ιωνί επόμενο βήμα. Αναφερόμενο ο κ. Μούλτερ στο άρθρο 23, όπω μα είπε και ο ίδιο στην ε, παρέμβασή του, ο κ. Μούλτερ θεωρεί ότι ε, για την επιτήρηση των συνόρων μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα χερσαία σύνορα ε, χωρίς κανένα πρόβλημα στο Eurosur. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία ε, Ξένια Γεωργιάδου ή ο κύριος ε, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης από πλευράς Κυπριακής Προεδρίας. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, good afternoon, Chair. Um... Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Η Κυπριακή Προεδρία θα ήθελε καταρχάς να συγχαρεί τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο έκθεσης και θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι η θέσπιση της Eurosur μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2013 παραμένει μια ισχυρότατη προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. μετά από όλες τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μάλιστα τον Ιούνιο του 2011. Για το λόγο αυτό και βασισμένη στην πρόοδο που επιτεύχθηκε υπό την Δανική Προεδρία, η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται να ε, συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για τον κανονισμό αυτό και στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας θα είναι μάλλον η τελευταία φορά όπου θα εξετάσουμε το σημείο αυτό σε επίπεδο ομάδων εργασία, και μετά θα το φέρουμε σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο στι επόμενε εβδομάδε υπολογίζουμε. Η Προεδρία ελπίζει οι διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με, για μια συμφωνία σε επίπεδο πρώτη ανάγνωση, να διεξαχθούν και να περατωθούν όσο δυνατόν ε, συντομότερα ευκταίων το τέλο του χρόνου. Το σχέδιο έκθεση του κυρίου Μάλντερ πιστεύουμε ότι είναι μια εξαιρετική βάση για περαιτέρω δουλειά και πραγματικά υπομονούμε να λάβουμε τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν ε, στα πλαίσια του σχεδίου έκθεσης. Η Κυπριακή Προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Μάλντερ για τη συνεργασία του και η συνεργασία αυτή ελπίζουμε να οδηγήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε μια ικανοποιητική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Ε, εδώ Σημειώσαμε ορισμένους που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Αρχίζουμε με τον κύριο Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρου του ΕΛΚ και εκ μέρου του κυρίου Σκούρια, του σκιώδου συζητητή του ΕΛΚ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μούλτερ για την έκθεση αυτή, για το σχέδιο έκθεση. Το ΕΛΚ καλωσορίζει την έκθεση αυτή και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε με τις ε, θέσει που υιοθετούνται από τον κύριο Μούλτερ. Επίσης, συμφωνούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα στο ότι στόχος του Eurosur θα, οι στόχοι του Eurosur θα πρέπει επίσης να ε, συμπεριλαμβάνουν και το να σωθούν ζωές στη Μεσόγειο και στις θαλάσσιες ζώνες. Πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση των εξωτερικών συνόρων μας και η ενίσχυσή τους έχει άμεση σχέση με το να σώσουμε ζωές, διότι η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων σημαίνει παρακολούθησή τους όλων των συνόρων και αυτό είναι ο μοναδικό τρόπος που ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε ζωές. Για μας λοιπόν η Eurosur είναι ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί καμία ζωή στη Μεσόγειο ή σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια ζώνη της ε, Ένωση. Δύο συγκεκριμένα σημεία θέλω να θίξω, ε, βασισμένοι στην, στο σχέδιο εκθέσης του κυρίου Μούλτερ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Καταρχάς, η ισχυρή υποστήριξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Πιστεύουμε ότι αυτή η άποψη της έκθεσης πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και φυσικά συμμεριζόμαστε τη θέση του κυρίου Μούλτερ. Όπως ο κύριος Μούλτερ και εμείς πιστεύουμε ότι η Eurosur για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν αποδοτικότερα χρειάζεται κάπως να συμπεριλάβει με πρακτικό και συμπαγή τρόπο τις τρίτες χώρες. Μετά, το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τις περιοχές πρώτων συνόρων. Και εδώ θα ήθελα μία διευκρίνηση, μάλλον. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Μούλτερ λέει ότι όταν συμπεριλαμβάνουμε τα συνοριακά περάσματα και τα αεροδρόμια, ότι ενώ αυτό είναι αποδεκτό για εκείνον, πιστεύει ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία. Θα ήθελα λοιπόν να ε, μου ξεκαθαριστεί εάν αυτό θα συμπεριλάβει και τις ε, θαλάσσιες περιοχές, διότι εμείς πιστεύουμε ότι οι περιοχές αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν άμεσα και δεν εννοώ μόνο τις ε, θαλάσσιες ζώνες που υπόκειται στην ε, αρμοδιότητα των ε, εκάστοτε των ανταπημέρους κρατών μελών, αλλά και οι θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες υπερβαίνουν τις ε, περιοχές που έχουν αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι αυτές οι ζώνες θα πρέπει να συμπεριληφθούν άμεσα στη δικαιοδοσία της Eurosur προς επιτήρηση. Ίσως λοιπόν ο κύριος Μούλντερ θα επιθυμούσε να μας το αποσαφηνίσει περισσότερο το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λούτφορντ. Μάλιστα, συγγνώμη που επεμβαίνω ξανά, Πρόεδρε, που πετάγομαι τόσο συχνά αυτό το απόγευμα. Και πάλι θίγω το θέμα από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θέλω να θεωρηθεί αυτό κάποια ειδική αναφορά. Όμως, ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που το Συμβούλιο και ο συνάδελφος Μούλτερ προτείνουν από κοινού τη δημιουργία διατάξεων, ειδικών ε, διατάξεων για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι ένα σημείο φυσικά. Κατανοώ απόλυτα το επιχείρημα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει τα περιθώρια να διαλέξει εκείνο τι προτιμά. Πράγματι, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει, ε, ένα, έχει μεγάλη δυνατότητα επιτήρησης, θαλάσσιας επιτήρησης και θα μπορούσε να ε, εντοπίσει λοιπόν τα σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο και να σώσει ζωέ στη θάλασσα. Υπάρχει όμω μια ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στο κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο και στο κείμενο που προτείνει ο κύριο Μούλτερ. Και ελπίζω να καταφέρω να πείσω τον κύριο Μούλτερ να κοιτάξει με θετικό βλέμμα τις προτάσεις και το Συμβούλιο φυσικά για το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει όχι μόνο με πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες, το Ηνωμένο ε, Βασίλειο και την Ιρλανδία, διμερείς λοιπόν συμφωνίες μεταξύ αυτών και ενός περισσότερων κράτη-μέλη, αλλά ακόμα παραπέρα να υπάρχουν, να, να υπάρχουν τέτοιε συμφωνίε που να αφορούν και τι γειτονικέ τρίτε χώρε. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αναμειχθεί σε συνεργασία ε, κρατών μελών και γειτονικών χωρών που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Και παίρνω αφορμή από τα λόγια του κυρίου Μπουσουτήλ για ισχυρή στενή συνεργασία ανάμεσα σε γειτονικέ χώρε. για να πω ότι εάν τα περιφερειακά δίκτυα δημιουργηθούν και τα δίκτυα αυτά συμπεριλαμβάνουν και κρατημέλη και μη κρατημέλη. Θα μου φαινόταν παράλογο να μην αφήσετε το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε αυτά τα δίκτυα, γιατί ε, του επιτρέπεται να, να ε, συνεργάζεται μόνο με κρατημέλη και όχι με τρίτες χώρες. Εγώ θα ε, συμπλήρωνα μία τροπολογία που θα καθρεφτίζει τα σχόλια και τις απόψεις στο σημείο αυτό, συνάδοντας βέβαια με την πρόταση του Συμβουλίου. Θα τον πιέσω τον κύριο Μούλτερ και προσωπικά για αυτό. Πιστεύω όμως ότι πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμμετάσχει βασισμένο στην, ε, στο, στην εύρυθμη λειτουργικότητα Πράγματι, είναι πολύ λογικό να επιτρέψετε στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε ένα ευρύτερο δίκτυο, περιφερειακό δίκτυο που συμπεριλαμβάνει και τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ πολύ τον κύριο Μούλντερ και να τον συγχαρώ για την εξαιρετική έκθεσή του. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες σας για τον κίνδυνο ζώων στη θάλασσα και την προστασία δεδομένων. Φαίνονται ξεκάθαρα στην έκθεσή σας. Τώρα για το αν η προστασία δεδομένων θα έχει το δικό της ε, αφιερωμένο άρθρο, είναι κάτι που εμείς το στηρίζουμε απόλυτα. Επίσης αναφέρατε το θέμα της ε, ευθύνης στις θαλάσσιες διασώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ένα σκάφος σε κίνδυνο στη θάλασσα είναι ένα πράγμα. Το να το βοηθήσει είναι κάτι άλλο όμω, είναι κάτι παραπάνω. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Θα θέλαμε να κάνουμε μερικές προσθήκες. Για παράδειγμα, την ανάγκη που βλέπουμε εμεί για ένα ημερολόγιο καταστρώματος για πληροφορίες που θα χρησιμοποιούνται σε ανταλλαγή με τα κράτη-μέλη. Μετά όσον αφορά τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ την Επιτροπή. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τις τρίτες χώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό είναι αναγκαίο. Γιατί είναι αναγκαία η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Ε, λέει εδώ ο κανονισμός ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να συλλέγονται. Αν συλλέγονται όμως γιατί να ανταλλάσσονται με τρίτε χώρε. Θα ήθελα μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Επίση, όσον αφορά το ποιο θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την Eurosur. Η Ευρωπόλ θα έχει πρόσβαση, Άλλε υπηρεσίε θα έχουν πρόσβαση. Υπάρχει ένα κατάλογο, είναι ανοιχτό, είναι κλειστό. Αυτό θα θέλαμε να μάθουμε. Ο κύριος Δεμέρη επίσης ανέφερε στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για το θέμα αυτό ότι η τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι πάντα αποδοτική, δεν, είναι, δεν έχει μαγικό ραβδί και κοστίζει και αρκετά. Τώρα, υπάρχει αυτό εδώ που σας δείχνω, υπάρχει αυτή η μελέτη ενός γερμανικού ιδρύματος που ασχολήθηκε με το κόστος που επιφέρει η Eurosur. Έγινε μια ανεξάρτητη έρευνα η οποία λοιπόν κατέληξε στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκτιμά το σύνολο του κόστου. Εκτιμά μικρότερο κόστος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή εκτιμά ότι το κέντρο εθνικού συντονισμού θα κοστίσει 99,6 εκατομμύρια ευρώ. Όμω, στην πραγματικότητα, τα κράτη-μέλη υπολογίζουν 105 εκατομμύρια ευρώ για το 2011 ως το 2013. Επίσης υπάρχουν επιπλέον υπάρχει ένα δις 200 εκατομμύρια για το μέχρι το 2020, το οποίο θα δοθεί και συνολικά φτάνουμε σε πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει εκτιμήσει η Επιτροπή. Μετά, σε άλλους τομείς, η, η Κομισιόν κάνει λόγο για εκτίμηση 129 εκατομμυρίων ευρώ. Η Frontex όμως υπολογίζει 20 εκατομμύρια παραπάνω μέχρι το 2013, εκτός από αυτών 132 εκατομμύρια ευρώ για, τον τομέ... για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανάμεσα στο 2014 και στο 2020. Γι' αυτό λοιπόν μας φέρνει πιο κοντά στα 152 εκατομμύρια. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό λοιπόν ανάμεσα στις δύο εκτιμήσεις. Επίσης βλέπουμε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις, ε, στα εργαλεία παρακολούθησης γίνεται αναφορά από την Επιτροπή για 29,6 εκατομμύρια, αλλά στην πραγματικότητα το κόστος, ε, το, που έχει δαπανηθεί, ε, το ποσό που έχει δαπανηθεί είναι 35 εκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο. Αν το, αν το αθροίσουμε αυτό τα τελευταία 10 χρόνια, και προσθέσουμε σε αυτό και τις έρευνες για, ε, και έρευνα και ανάπτυξη, τότε θα δούμε ότι το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Και που καταλήγουμε, δεν καταλήγουμε σε... Καταλήγουμε στα 350 εκατομμύρια ευρώ και είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Έπειτα, τα δίκτυα με τις τρίτες χώρες. Η μελέτη δείχνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στις εκτιμήσεις της Κομισιόν και στις εκτιμήσεις ύψους 98 εκατομμυρίων ευρώ, ευρώ της έρευνας αυτής. καθώς επίσης και για το, πρόγραμμα, για το, το κόστος μετάβασης από το ΣΥΣ στο ΣΥΣ 2 και το κόστος ε, των ε, τρίτων ε, χωρών συμμετοχή, της συμμετοχής του στη Eurosur. Με τα χαράς να στείλω την έρευνα σε όλους σας. Είναι μια ανεξάρτητη έρευνα, όπως είπα. έχουμε λοιπόν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 38,7 εκατομμύρια ευρώ και τις εκτιμήσεις της ανεξάρτητης μελέτης 873. Η Επιτροπή ίσως θα μπορούσε να κοιτάξει τα νούμερα αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες, να τα εξετάσει. Εγώ προσωπικά όταν ε, διάβασα την έρευνα τη θεώρησα αρκετά πιστική και πιστεύω πως πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι αυτά τα κονδύλια είναι ένα τεράστιο ποσό και ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο κρίσης που ζούμε. Φτάνουμε σχεδόν στα 900 Φυσικά θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας μικρές προσθήκες, όμως το ζήτημα του κόστους από το ζήτημα του κόστου προκύπτει μια ερώτηση. Γιατί είναι απαραίτητη η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τρίτε χώρε. Και αυτό θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ε, ευχαριστώ. Συνάδελφο Κολίνα. Ο κύριος Γιακολίνο, εγώ θεωρώ απόλυτα ε, συμπατή τη θέση του κυρίου Μιούλντερ με τις ε, αρχές που διέπουν το όλο ντοσιέ. Τώρα η συνάδελφος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο κόστος ωφέλεια. Παρατηρήσεις με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οι, τροπολο... οι τροπολογίες 13 και 15 προβλέπουν στο 13 όλα τα κράτη-μέλη να αφορά σε όλα τα κράτη-μέλη. Το μέτρο ασχέτως που βρίσκονται. Πρέπει όμως να το συνδυάσουμε και με το 15 που σχετικά με τα κέντρα συντονισμού προβλέπει και μία ειδική αρμοδιότητα επιτήρησης των συνόρων. Εγώ θεωρώ ότι είναι ασύμβατες αυτές οι δύο δράσεις και θα δημιουργούσαν δυσκολίες. Θα ήθελα να το σκεφτεί αυτό και ο εισηγητής και η Κομισιόν. Ο στόχος της Ευρωσούρ είναι να ενισχύσει τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα και αυτό θα αποτελούσε και την προστιθέμενη αξία όπως επίσης ε, και την ε, προστασία απελπισμένων μεταναστών μέσα στη Μεσόγειο. Το ποιοτικό άλμα σε όλη αυτή την ιστορία είναι οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Θα έλεγα λοιπόν στον κύριο Μούλτερ να εξετάσει και αυτή την εναλλακτική λύση στην τροπολογία 42 ακριβώς όταν αναφέρεται για την προστασία της ζωής των μεταναστών σε διμερείς συμφωνίες για την καταπολέμηση της εγκληματικότητα και ξέρετε ότι η λαθρομετανάστευση πολλές φορές βρίσκεται στα χέρια της εγκληματικότητα. Λέει λοιπόν ότι χρειάζονται πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Αυτό θα ήταν ένα ποιοτικό άλμα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε μέσα από νόμιμη μετανάστευση να αντιπαρατεθούμε στο φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης. Η κυρία Μάκεντάιρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλη τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε για τους συγκεκριμένους στόχους του εγχειρήματος. Θα αποτραπεί η τραγική απώλεια ανθρωπίνων ζώων στη Μεσόγειο. Ε, και ελπίζουμε να μην επαναληφθούν τραγωδίες του παρελθόντος με τα νέα μέτρα. Θα τον ευχαριστούμε επίσης για τη συνεργασία μας στις συσκέψεις των σχεδόν εισήγητων. Έχει ήδη συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσης κάποια από τα πράγματα που του ζητήσαμε. Ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερο και είναι το πρώτο από τα τρία που θα θίξω είναι το εξή. η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Ο εισηγητή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχαν την ευγενή καλοσύνη να επεκταθούν λίγο ε, σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό προβλέπουν θα μπορούσε ενδεχομένω να συμμετάσχει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Η Βαρόνι Λάτφορντ αναφέρθηκε σε αυτό ε, το θέμα, στα πολλά που έχει να προσφέρει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και στην επιθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να προσφέρει, στο, να συμμετάσχει στο όλο εγχείρημα. Θα ήταν κρίμα ε, να μην αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό που μας προσφέρει. Ε, γιατί επιλέξατε να υποβάλλετε την τροπολογία επί τη βάση του άρθρου 17 και όχι του 18. Υπάρχει κάποιος ε, λόγος για την επιλογή που κάνατε που σχετίζεται ενδεχομένως με τη δική σας άποψη περί ενδεχόμενης συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Δεύτερο σημείο θα ήθελα να καταγραφεί η ανησυχία μου, όπως ανέφερε και η προλαλήσασα, ε, ως προς ε, το κόστος ε, που συνεπάγεται αυτό το εγχείρημα. Οι τεχνικές προκλήσεις είναι πελώριες στο εγχείρημα αυτό και δεν γνωρίζω εγώ κανένα πληροφοριακό σύστημα που να συνεπάγεται τόσο μεγάλο κόστος ε, όσο αυτό σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δηλαδή θα πρέπει να μετριάσουμε λίγο τις εντυπώσεις που δημιουργούνται ε, και θα ήθελα να με διαβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούν να υποστηρίξουν το κονδύλι ε, που προτείνεται. Με ποιο τρόπο θα κρατήσουμε υπό έλεγχο το κόστος του εγχειρήματος θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει περαιτέρω. Τρίτον, και απευθύνομαι τόσο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής όσο και στον εισηγήτη και ε, σχετίζεται με το άρθρο 15. Με ανησυχεί διότι ε, εδώ εξετάζουμε ζητήματα εθνικής ασφάλειας ε, που προφανέστατα υπάγονται αμυγός στην εθνική αρμοδιότητα. Γιατί λοιπόν προβλέπει τις αντιδράσεις του κράτους μέλους η Επιτροπή μέσα στην πρότασή της ε, σε σχέση με ε, γιατί προβλέπει τις αντιδράσεις του κράτους μέλους σε σχέση ε, με τις δράσεις του Frontex μήπως παρεμβαίνουμε στα χωράφια της εθνικής ασφάλειας αυτό ήταν το τρίτο ερώτημά μου και ευχαριστώ και την Επιτροπή και τον κύριο Μόλτερ ευχαριστούμε κύριε Μπρόνς ήρθε η σειρά σας ευχαριστώ πρόεδρε όλα τα βήματα πρέπει να γίνουν για να αποφευθούν οι θάνατοι πάνω στα φουσκωτά στη Μεσόγειο πρέπει να γίνουν, όντως. Και είμαι ε, σίγουρος ότι η συγητής θα συμβάλλει ότι μπορεί ε, σε αυτό το θέμα. Όμως, ε, οποιαδήποτε αποτυχία να σώσουμε ε, ζωές ε, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ε, γίνει αποδεκτή. Για να βρούμε τη λύση όμως δεν πρέπει να εξετάσουμε γιατί διακινδυνεύουν τη δική τους τη ζωή των συντρόφων τους ακόμη και των παιδιών τους αυτοί οι μετανάστες σε ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Αν αποφύγουν αυτό το κίνδυνο του να βουλιάξει η βάρκα και να πνιγούν και βγουν στη στεριά ή θα πάρουν άσυλο ή θα απορριφθεί το αίτημά τους αλλά θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ούτως ή άλλως. Η υποχρέωση υποδοχής ετούντων άσυλο που εισήλθαν παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από ανθρώπινα μυαλά. Δεν είναι θέσφατο πράγμα και μπορεί ένα ανθρώπινο μυαλό να τροποποιήσει αυτή την υποχρέωση καταργώντας έτσι το κίνητρο που έχουν οι μετανάστες αυτοί που διακινδυνεύουν ξαναλέω και τη δική τους τη ζωή και αλωνών για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέτοντας ένα τέρμα σε, αυτά, σε αυτή την επικίνδυνη διαδικασία. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μπρόνς. Ε, θα είδατε ότι όσο πλησιάζει η ώρα της ψηφοφορίας ε, που έχει προβλεφθεί για τις 6.30 γεμίζει και η αίθουσα. Ναι, ήρθε η ώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει σε ερωτήσεις ε, που τις απίφθηναν τα μέλη της Επιτροπής. Ε, παρακαλώ η Επιτροπή και ε, θα κλείσει τη συζήτηση ο εισηγητής μας ο κύριος Μούλτερ. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα σχόλια. Δεν έχουμε χρόνο και άρα θα είμαι κι εγώ σύντομος. Ε, δεν θα μπορέσω όμως άμεσα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις ως εκ τούτου. Αναφερθήκατε στην γενικότερη κατάσταση της χρήση των πληροφοριών. Ε, σας παραπέμπω στο άρθρο 11, εδάφιο 3, όπου ρητά συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα επιτήρησης ε, αερολιμένων ε, και ελέγχων των σημείων διέλευσης των χερσαίων συνόρων για να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα ως προς τις ασφάλειες τις πληροφορίες ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσικό επόμενο των αντίστοιχων κινήσεων που έχουν γίνει για τα ε, θαλάσσια σύνορα, παραδείγματο χάρη. Ω προ τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε και αν αυτό θα συνδυαστεί με τη συμμετοχή ή όχι ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ιρλανδία, Δεν μας δημιουργεί πρόβλημα αυτό καθεαυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως αντίθετα θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρο σε σχέση με τις προθέσεις του προτείνει συνεργασία στην Μεσόγειο, διότι ε, τώρα συνεργάζονται με το δίκτυο Seahorse της Μεσογείου ή ε, μιλάμε για ε, χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου ή όχι, δεν θέλω να εισέλθω σε λεπτομέρειες διότι είναι λεπτό πολιτικό ζήτημα αυτό. Ε, θα μπορούσε να, κανείς να αμφισβητήσει την προσθέμενη αξία της ε, συμμετοχής ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Απ' την άλλη όμως θέλουμε τον Οκτώβρη του 2013 να είναι πλήρως λειτουργικά τα συστήματα. Θέλουμε να χαθούμε μέσα σε συζητήσεις τέτοιου τύπου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα καλύψει και τον Ατλαντικό. Ε, αυτό αναρωτιόμαστε, αλλά δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους ε, και να ε, διαπιστώσουμε από πολιτική ε, σκοπιά τι είναι πλέον επιθυμητό από πλευρά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν είναι σίγουρα δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να ασχολείται με τέτοια πολιτικά ζητήματα. Ένα λεπτάκι για να μην ξεχάσω κάτι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάβασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την μελέτη που ονομάζεται Borderline που ζήτησε η ομάδα των Πρασίων και στην οποία αναφερθήκατε. έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια για να κατανοηθεί το όλο εγχείρημα του Eurosur σε όλες του τις διαστάσεις. Ε, βεβαίως ε, θα το εκτιμούσαμε αν οι συντάκτες ε, αυτής της μελέτης θα είχαν κάνει μία φορά μία προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσουμε μία απάντηση για κάποιες υπόνοιες της έκθεσης σε σχέση με το κόστος ε, του Eurosur γιατί ορισμένες, απο, ορισμένοι ισχυρισμοί είναι απλώς εσφαλμένοι. Ε, μιλήσαμε επίσης για μια δεκαετή ε, περίοδο, αξιολόγηση του κόστους δηλαδή για μια δεκαετή περίοδο και δεν έχει συμπεριληφθεί αυτό στην αξιολόγηση αντικτύπου. Κοιτάξτε, το κόστος δημιουργίας μιας υποδομής, θα μιλάμε για δίκτυο ή για συγκεκριμένη υπηρεσία, είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα είναι το κόστος συντήρησης της υποδομής ε, ή του δικτύου. Όταν μιλάμε με την βιομηχανία διαπιστώνουμε ότι μας περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Δηλαδή η βιομηχανία εκτίμησε ότι η εκκίνηση και μόνο του δικτύου ε, αξίζει 10 εκατομμύρια τουλάχιστον. Ε, και η Frontex ε, κατάφερε να επιτύχει την θέσπιση με 1,5 εκατομμύριο μόνο του συστήματος, διότι θα χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο με κωδικοποίηση ασφαλείας των δεδομένων και έτσι με 1,5 εκατομμύριο να πτήσουμε αυτό το δίκτυο και διασυνδέεται με όλα τα υπόλοιπα. Ε, και θα χρειαστεί άλλο 1,5 εκατομμύριο για τα επόμενα 12 ε, κράτη-μέλη, πέρα από τα 6 που θα το εφαρμόσουν δηλαδή σε μια πρώτη φάση εξού και τα διάφορα ποσά που βλέπετε στην αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού. Όντως αληθεύει ότι η εκτίμηση του κόστους είναι μάλλον χαμηλότερη του πραγματικού, αλλά ε, πρέπει να γνωρίζετε ότι επιλέγουμε πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αξιολογήσεις αντικτύπου την ε, λιγότερο ε, πώς να σας πω, περιοριστική λύση. Δηλαδή, ε, αποφασίσαμε ότι ε, δεν θα έχουμε command and control. Θα έχουμε απλή χρήση του συστήματος Eurosur. Θα έχουμε ελέγχους στα σύνορα και όχι συνολικότερη επιτήρηση και των θαλασσίων σύνορων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και άλλες εναλλακτικέ λύσεις που όμως αυξάνουν ε, έτσι περαιτέρω το κόστος. Θα μπορούσα να σας δώσω και περισσότερα παραδείγματα για να στηρίξω τη θέση θέση μου, αλλά πολύ φοβούμαι ότι ε, δεν έχουμε χρόνο. Εάν αντίθετα κάποιος ενδιαφέρεται όλος ιδιαίτερο για το θέμα του κόστους, είμαι στη διάθεσή σας. Ήθελα μόνο κλείνοντα να σας πω πως ε, από αυτά που έχουμε δει δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα, αλλά από ό,τι φαίνεται το κόστος του Eurosur ε, είναι χαμηλότερο του εκτιμόμενου Ήμασταν ε, επίσης ε, γενναιόδοροι μάλλον σε σχέση με τα ποσά που θα λάβει ο Frontex, δηλαδή δεν έχουμε ε, τόσο μεγάλο πρόβλημα με τα ποσά, αλλά έχουμε πρόβλημα με το Frontex, δηλαδή ποια θα είναι η πηγή των κονδυλίων, αλλά αυτό είναι ξεχωριστή συζήτηση. Τι άλλο αναφέρθηκε. Ο κύριος Τζακολίνο. Μας ρώτησε αν ε, στις συμφωνίες ε, με τρίτες χώρες, αν εννοήσα ορθώς, ε, ρωτήσατε αν θα πρέπει να υπάρχει μια πρότυπη συμφωνία, μία και μόνο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι υπόλοιπες τρίτες χώρες ή αν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μια πληθώρα διμερών συμφωνιών. προκρίναμε τη δεύτερη λύση. Πρόεδρε, να τελειώσω την πρότασή μου. για τον εξή λόγο διάφορες ε, τέτοιες ε, συμφωνίες προϋπάρχουν, διμερείς εννοούμε, και άρα δεν ε, χρειάζεται να ξεκινήσουμε και πάλι νέες διαπραγματεύσεις, διότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε και τον κύριο Μόλτερ για να κλείσει η συζήτηση. Παρακαλώ, δείτε και το ρολόι, γιατί έχουμε αρκετές ψηφοφορίες. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, Πρόεδρο. Καταρχάς, χαίρομαι που έχω την υποστήριξη των περισσότερων. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω πολύ λακωνικά για τα σχόλια που διατυπώθηκαν. Καταρχάς για αυτό που είπε ο κύριο Μπουσουτήλ, ναι, τα, ε, οι θαλάσσιε περιοχές μπορούν να συμπεριληφθούν. Όχι απαραίτητα μόνο όταν χρειάζεται, αλλά μπορούμε να το κοιτάξουμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τι ανησυχίε τη κυρίας Λάτφορντ, για την συμμετοχή του ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν το θεωρούμε ιδιαίτερη περίπτωση. Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό θα επωφελήσει έτσι κι αλλιώς όλους μας. Ε, θα κοιτάξουμε την διατύπωση της ανταλλαγής πληροφοριών ε, υπό την προϋπόθεση όμως να έχουν όφελος και τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Μπορούμε να το συζητήσουμε όμως αυτό. Κυρία Κέλλερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, ε, ε, για για την υποστήριξή σας. Από την αρχή ζήτησα και εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου απαντήσει αν είναι επαρκή ε, οι ε, διατάξεις του προϋπολογισμού. Όχι, δεν είναι και γι' αυτό χρειάζεται να εισαχθούν στο νέο σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχω κάποιε ενδείξει όμως ε, και σύμφωνα με αυτέ, το κόστο αναμένεται να είναι υψηλότερο από όσο αναμέναμε. Κύριε Γιακολίνο τώρα, νομίζω πως ε, εισήγαγα την ε, τροπολογία διότι είναι βασισμένη στο Σέγγεν. Το Σέγγεν είναι υπεύθυνο για όλα τα μέλη του, ανεξαρτήτως εξωτερικών ή όχι συνόρων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από την αρχή να συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες. Κυρία Μάκιντάιρ, δεν μπορώ να σας πω τι χρειάζεται στην περίπτωση του ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορώ να σας πω ότι αφήνω ανοιχτό τον δεχόμενο διμερών συμφωνιών με το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει η δυνατότητα και πρέπει να, διαπραγματευ... να γίνουν οι αναγκαίε διαπραγματεύσεις γι' αυτό. Κύριε Μπρόντ, συμφωνώ ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Ή αυτό αν δούμε τις περιπτώσεις των ανθρώπων που ρισκάρουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο για να εισέλθουν, είναι προς το, είναι προς το συμφέρον όλων μας και των γειτονικών κρατών και των κρατών μελών να υπάρξει ευθύνη πληροφόρησης, έγκαιρης πληροφόρησης για τις μετακινήσεις των προσφύγων για να μπορέσουμε λοιπόν να αναλάβουμε δράση πρωτού είναι αργά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μούλτερ και για την προσπάθεια αυτή περίληψης. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι η Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στο μεσημέρι. Η συζήτηση των τροπολογιών στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προβλέπεται ε, για τις 10 και 10 Οκτωβρίου και η ψήφος ε, προσανατολισμού θα λάβει χώρα στο τέλος Νοέμβρη. Αφού λοιπόν αν σας είπα αυτές τις ανακοινώσεις, τώρα προχωρούμε στην ψηφοφορία. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μισή ώρα. Γι' αυτό συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Διότι έχουμε ένα σημείο ακόμα στην ημερησία διάταξη, αφού ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία για μισή ώρα. Αρχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. πρόταση για το εφαρμοστέο δίκαιο για την ε, πρόταση της συναδέλφου Εύελιν Γκέμπχαρτ. Αρχίζουμε με τις τροπολογίες. Αν είστε έτοιμοι. Σημείο 8 της ημερήσιας δίδαξης. Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Υιοθετη... Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 11. Για την 11 ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 28 ψήφοι υπέρ, 18 ε, κατά. Μία αποχή εγκρίνεται.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 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Όχι, παραμένει, παραμένει η 35. Α, όχι, όχι, πέρασε, πέρασε η προηγούμενη. Οκ, okay. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίθηκε λόγω των αποχών δηλαδή. Λοιπόν, οι εποχές ήταν παραπάνω από τα ναι και από τα όχι. Λοιπόν, 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε για την 38 αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 22... Τι έγινε? Πού πήγε η οθόνη? Δεν φαίνεται πια. Τι έγινε ο τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Να ξαναψηφίσουμε, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, για την 38 ελέγχουμε και αρχίζει ψηφοφορία τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ 22 κατά απορρίπτεται με 7 αποχές. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20... Συγγνώμη, συγγνώμη, πάμε στα εκτιμώντας τώρα. Λοιπόν, 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, είδα παραπάνω χέρια, είδα παραπάνω ναι, από ότι όχι. Να ελέγξουμε για την 28. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Λοιπόν, πάμε στην τροπολογία 1, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 2 και οι 29 είναι ίδιες, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε συνολικά το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά λοιπόν αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Ωραία, τώρα κλείνουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. 45 υπέρ 4 κατά 0 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Γκέπχαρτ. Προχωράμε λοιπόν. Πάμε τώρα στις αποφάσεις σχετικά με τον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχειρημένων συντρόφων.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 κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 εδώ έχουμε ένα συμβιβασμό για την 17 και την 35 ψηφίζουμε έχετε το κείμενο για τον συμβιβασμό δεν το έχετε να σας το διαβάσω. Λέει τα Α, το, έχετε. Εάν ε, το έχετε όλοι λοιπόν. Το έχετε όλοι. Είστε σύμφωνοι να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. Όχι, ναι. Ας το διαβάσουμε. Έτσι για τα πρακτικά. Λοιπόν, το κείμενο λέει η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί προτέρως, οι σύντροφοι μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο εάν, εφόσον ο νόμος του ε, κράτους ε, διαμονής αναγνωρίζει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 κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 30, 31 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν εκτιμώντας 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτός μικροφώνου. Ψηφίσαμε. Τροπολογία προς τροπολογία. Και υπήρξε συνένεση. Πέντε υπέρ. Τέσσερα, τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέλικη ψηφοφορία στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 46 υπέρ, 3 ε, κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Κάρσμαν και σας ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρτ που εκπροσωπήσατε τον συνάδελφο σε αυτήν την έκθεση. Πάμε τώρα στην τρίτη ψηφοφορία. Είναι μία πρόταση απόφασης για το ευρωπαϊκό... σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Ελπίζω να μην έκανα λάθος. Πρόκειται εδώ περί του συμβιβασμού που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν. Πρόκειται λοιπόν για ένα συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο σημαίνει ότι ψηφίζουμε στο συμβιβαστικό κείμενο και μετά στην τροποποίηση του κειμένου. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το τελικό κείμενο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίες. 45 υπέρ 2 κατά 2 αποχές. Ευχαριστώ κυρία Παπαδοπούλου για τον συμβιβασμό. Τώρα. Γίνονται ευκολότερα τα πράγματα. Ξέρετε τι καταφέραμε, 30 τόσες, σχεδόν 40 σελίδες τροπολογίες γλιτώνουμε. Τα γλιτώσαμε. Τώρα θα ψηφίσουμε. Όχι, δεν τα λέω καλά. Κι όμως, Ψηφίζουμε τώρα για τις τροπολογίες του, για τον προπολογισμό. Ο Σαλβατόρε Γιακολίνο είναι ο εισηγητής, ο οποίος είναι, ένας, ε, είναι τακτικότατος στο θέμα των ε, τροπολογιών. Την 56 ε, και την 70... 56, 70. Έχει αποσυρθεί η 5670. Όχι η 56 και 70, η 5670. Έσβησε το μικρόφωνο του Πρόεδρου στο μεταξύ. Δεν ακούγεται. Getting started, Θα αρχίσουμε. Παρακαλώ να συγκεντρωθείτε 5613 υπέρ. Κατά. Αποχές 5614 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 56-15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56-16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56-17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56-18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56-19 είναι συμβατή, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56-20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5681 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5622 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5623 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5601 υπέρ, κατά αποχές να το ελέγξουμε δεν είναι καθαρό λοιπόν 56-0 να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία παρακαλώ άρχισε η ψηφοφορία ψηφίσατε ε, πέρας ψηφοφορίας κλείνουμε κλείνουμε Η 26 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. Ως εκ τούτου 56-26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56-02 υπέρ κατά αποχές Θα έλεγα ότι αν έχουμε την ίδια πλειοψηφία με προηγουμένως εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. 5602. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 26-24 το σκορ. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει πλειοψηφία λοιπόν. Ναι, όχι. 56-28. Ναι, όχι. 56-28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56-29 υπέρ. Κατά αποχές 5631 56-31 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. 56-31, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. 22-28 το σκορ απορρίπτεται. 56-32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56-32. 33, 56-33, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56-34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56-35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. 5636. είναι ο προεδρο κατα αποχέ αποχές εγκρίνεται 56-37 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται 38 ενωντας 5638 56-38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5603 υπέρ. Οι 40 και 41, 56 ε, μπροστά γιατί είναι ίδιες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 56-42. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56-04 υπέρ και η 43 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε, να ελέγξουμε, γιατί είναι ίδιες. Η 04 και η 43, αρχίζει η ψηφοφορία. Ελέγχουμε, πέρας ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 6 κατά.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 κατά απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 07 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να το ελέγξουμε Ελέγχουμε λοιπόν για την 07. Αρχίζει η ψηφοφορία. 07, 07, ναι. Πέρας ψηφοφορίας. 26-24 εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64, 65 και 66 είναι ίδιες τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, η 56, 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε για την 69. Να το ελέγξουμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 26-21. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 71, την 5671, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 19-29, το σκορ απορρίπτεται. 08 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 να, ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 77 ελέγχουμε την 77 ηλεκτρονικά αρχής ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 19-28 απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές χρειάζεται έλεγχος για την 79 αρχίζει ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας 28-22 εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, συγγνώμη, συγγνώμη να το επαναλάβουμε, να το επαναλάβουμε το 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε εγκρίνεται τελική ψηφοφορία Τροπολογία 1 της voting list. Υπέρ. Στην τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Τροπολογία 2. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε, να ελέγξουμε το 1. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 1. Η ηλεκτρονικά. Αρχής ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. 21-29 το σκορ. Απορρίπτεται για τη 2 υπέρ κατά αποχές. Τώρα εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέρασε λοιπόν η τέσσερα, Η... Για την πέντε λοιπόν τώρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια κύριε Γιακολίνο. Λοιπόν, να, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πάλι εδώ έχουμε μία άσκηση συμβιβασμού. Σας ευχαριστώ κύριε Μούλντερ που κάνατε τη δουλειά, διότι μας ε, βοηθήσατε πολύ. Εάν ψηφίσουμε το συμβιβαστικό κείμενο, λοιπόν, υπέρ αυτού του συμβιβαστικού κειμένου, κατά αποχές εγκρίνεται. Και το τελικό κείμενο τώρα, υπέρ. Αρχίζει, συγγνώμη, ψηφοφορεί ηλεκτρονικά. 50 υπέρ, καμία, κανένας κατά καμία αποχή. Ομοφωνία, ομοφωνία για τη χρήση προδρόμων ουσιών εκρηκτικών υλών. Μπράβο κύριε Μιούλτερ, μπράβο. Ε? We're getting close to the end. Κουράγιο και πλησιάζουμε στο τέλος. Ε? The boast is there. The, the boat is there. Eh? How are you? Okay. You kindly requested to leave the room in silence. Παρακαλώ, αν μπορείτε αθόρυβα, ώστε δυνατόν πιο αθόρυβα γίνεται να φύγετε από την αίθουσα όσοι είναι να αποχωρήσετε για να περάσουμε εμείς την έκθεση κυρία Έντιτ Μπάουερ. Ένα λεπτάκι. Silence in the ranks. Ησυχία Dear colleagues, Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Λοιπόν, όσοι μείνατε στην αίθουσα ησυχία. Είναι το σημείο 13, προξενική προστασία για τους πολίτες της Ένωσης στο εξωτερικό. Η συγγήτρια είναι συνάδελφος κυρία Μπάουερ. Πρόκειται για την εξέταση των τροπολογιών στην πρόταση του Συμβουλίου. Έχουμε εμεί εδώ τις τροπολογίες. Έχουμε και την έκθεση. Θα ακούσουμε την κυρία Μπάουερ και μετά θα ολοκληρώσουν οι συνάδελφοι, όπως επίσης θα ολοκληρωθούν και οι εργασίες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, για τις ε, προτάσεις. 106 προτάσεις για, για συμβιβαστικές έχω λάβει, συν τις αρχικές τροπολογίες. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που τελικά δέχτηκαν τη γραμμή μου. Βέβαια υπάρχουν ακόμη μερικά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Για παράδειγμα το θέμα της προσωπικής εφαρμογής ε, των προξενικών διατάξεων είδαμε, διαπίστωσαν οι συνάδελφοι ότι στο αρχικό κείμενο δεν έχουμε πια τον όρο ε, συγγενής... Ε, οικογένεια κλπ. Ε, δεν τον έχουμε πια αυτόν τον όρο. Μας είπανε ότι η υπερρυθμιστικότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα. Δηλαδή, μέλη της οικογένειας που ζουν σε μία τρίτη χώρα θεωρούνται μέλη της οικογένειας μέχρι τα 21 έτη. Φανταστείτε εσείς Φανταστείτε τι γίνεται όταν μπορούμε να, να επέμβουμε και να σώσουμε ένα μέλος της οικογένειας που είναι 21 ετών και δεν μπορούμε να σώσουμε εκείνο που είναι 22. Οπότε μας είπανε μην ρυθμίσετε υπερβολικά το θέμα, διότι αν επιτόπου οι αρχές επιμένουν στη λεπτομέρεια της ε, νομοθεσίας, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ζημιά. Τι θα γίνει, θα αφήσουμε την αναφορά στο κείμενο ή θα σβήσουμε την ίδια την αναφορά. Οι τροπολογίες 47, 49, 55, 71, 85 επίσης δημιουργούν πρόβλημα διότι το εφαρμοστικό πεδίο αυτής της οδηγίας ε, θα αφορούσε και τους απάτριδες. Αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει έναν δεσμό μεταξύ της προξενικής προστασίας και της υπηκότητας ενός κράτους μέλους. αν στο προήμιο έχουμε την πρόταση της κυρίας Ανούτα. και καλύψουμε άτομα τα οποία δεν προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, δημιουργούμε πρόβλημα. Αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι ποιον θα καλύπτει η προξενική προστασία. Η νομική βάση τελικά τι είναι, ο συντονισμός. Εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε στο, στα όρια της εναρμόνισης, αλλά δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε νέες υποχρεώσεις ε, στα κράτη-μέλη. Η προξενική προστασία ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη. Παρακαλώ λοιπόν στους συναδέλφους να μην θελήσουν να επιβάλλουν νέες υποχρεώσεις, να μην ορίσουν νέες υποχρεώσεις πρέπει πάντα να παραμείνουμε μέσα στα επίπεδα του συντονισμού. Ορισμένοι συνάδελφοι και θα έπρεπε σε μία επόμενη φάση η εξωτερικές υπηρεσίες της Ένωσης ε, να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την ε, προξενική αρχή, την προστασία της προξενικής αρχής. Εγώ δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα ήθελα εγώ η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου να παίζει ένα ρόλο και έναν ρόλο κέντρου. Θα, έπρεπε, θα πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει την δυνατότητα να, ε, να επιλέγει μία προξενική αρχή. Εξού λοιπόν και οι τροπολογίες 75 και 76 δεν είναι δεν με βρίσκουν σύμφωνοι διότι αντιφάσκουν με την συνθήκη. Τώρα, δεύτερη, πρώτο άρθρο του 2, δεύτερη παράγραφος του 4, άρθρο 14, μας, βάζουν, μας θέτουν ορισμένες δυνατότητες συμβιβασμού και εμεί μπορούμε κάλλιστα να βρούμε συμβιβασμό για αυτά τα άρθρα. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθω σε επαφή και θα έρθω σε επαφή και με τους σκεώδεις εισηγητές, αλλά θα κοιτάξω να βρω συμβιβασμό για όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξωτερική της δουλειά. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Αλλά επιμένω στο ρόλο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μπορεί να είναι αποτελεσματική προξενική προστασία και να είναι και καλά συντονισμένη, θα πρέπει ο πολίτης να μπορεί να, να καρπούται πλήρως των δικαιωμάτων του στην προξενική προστασία βάσει των συνθήκων. Γι' αυτό και κατέθεσα εγώ τις τροπολογίες σε μία φάση κρίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικό συντονισμό και καταμερισμό ε, αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντονίζει τις προσπάθειες και δεν κάνω πίσω σε αυτό. Καταλαβαίνω εν μέρη το επιχείρημα της κυρίας Μπάουερ, αλλά έχω ένα πρόβλημα για τις αντιπροσωπείες. Είναι το θέμα του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών έτσι όπως αναφέρονται και στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ δεν έχω καμία εγγύηση στο κείμενο που εσείς μας ε, δίνετε εδώ ότι ένα ζευγάρι ομοφιλοφίλων θα το αντιμετωπίσει θα αντιμετωπιστεί ισότιμα από τη μία ή από την άλλη προξενική αρχή ενός κράτους μέλους και αυτό γιατί λείπει σχετική νομοθεσία σε ορισμένα κράτη-μέλη. Σίγουρα ξέρω ότι δεν ε, απέχουμε από τη συμφωνία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα θέμα καταμερισμού ευθυνών για, αυτό το, και για, αυτές τις πλευρές. Επίσης, κυρία εισηγήτρια, εσείς αφήνετε την προξενική βοήθεια στις διπλωματικές αρχές των κρατών μελών. Και γιατί δεν θέλετε να δώσετε ένα σημαντικότερο ρόλο στις αντιπροσωπείες της Ένωσης και να τις αναθέσετε και ε, και αρμοδιότητες. Αυτό θα ε, αυξήσει την σημασία, σημασία και το ρόλο των αντιπροσωπιών. Εμείς κοινοβούλιο είμαστε εδώ, οπότε όσο το δυνατόν, ε, όντας κοινοβούλιο, όσο πιο πολύ ενισχύουμε εμείς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τόσο το καλύτερο πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες θα μπορούσαμε έτσι να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα στην Ένωση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, αναθέτοντας την προξενική προστασία στις αντιπροσωπείες, ε, δεν θα έχουμε την εγγύηση ότι θα γίνονται σεβαστά, ή τα, σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να με διασφαλίσετε σχετικά με το θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω καμία εγγύηση, συγγνώμη, γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι πρεσβείες και τα προξενία των κρατών μελών εγγυώνται τα ίδια δικαιώματα στα ομοφιλόφιλα ζευγάρια και στα μέλη της οικογένειάς τους. Ποιος μου το εγγυάται εμένα αυτό. Όταν έχω εγώ εδώ το κείμενο δεν έχω την απόλυτη εγγύηση για μια τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζητώ σε ορισμένες ε, περιπτώσεις να αντιπροσωπεύει, να αντιπροσωπεύονται από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτήν την εγγύηση την έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη, όχι. Όταν βλέπω και ορισμένες συμπεριφορές ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών ε, έναντι των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για τέτοιου είδους ζητήματα πραγματικά τρέφω τεράστιους ε, φόβους. Κυρία Μπάουερ, δεν απέχουμε ε, στις θέσεις μας. Εγώ πιστεύω ότι συζητώντας θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη διασφάλιση. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ρεαλιστής, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο σύστημα ε, για τις αντιπροσωπείες και έναν ενισχυμένο ρόλο, αλλά πολλά πράγματα οι αντιπροσωπείες μπορούν να το κάνουν. Όταν έχουμε να κάνουμε με προξενία και πρεσβείες κρατών μελών που δεν έχουν στην νομοθεσία τους αυτή την ερμηνεία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η μόνη προσφυγή λοιπόν είναι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευέλικτος βέβαια, ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνατε, σας συγχαίρω και Είμαι στη διάθεσή σας να βοηθήσω για να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί κατά τη γνώμη μου μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ κύριε Μισελ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ε, θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν όχι, η Κομισιόν θέλει το λόγο. Όχι. Α, δεν είναι εδώ η Κομισιόν, ωραία. Το λόγο έχει και πάλι ο κύριος Μπάουερ, λέει ο πρόεδρος για την κυρία Μπάουερ. 19-20 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε. Κυρία Μπάουερ. Thank you uh, for the possibility to react. Uh. Ευχαριστώ που μας δίνετε, μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω και πάλι το λόγο μετά τις προτάσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους νωρίτερα ανέφερα ότι υπάρχει μια αντίφαση ε, στον ορισμό που δίνουμε για τα μέλη της οικογενείας. Στην οδηγία 38 υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος καλύπτει τα ζευγάρια των ομοφιλοφίλων αλλά ε, απ' την άλλη, ε, ε, αν συμπεριλάβουμε αυτόν τον ορισμό, έχει αυτό κινδύνους για άλλους, όπως η η υπήκοοι τρίτων χωρών άνω των, του 20, των 21 ετών. παρότι είναι ε, μέλη της οικογένειας. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό που έρχεται από αυτήν την οδηγία 38, αυτά τα άτομα δεν θα γίνονται δεκτά ως ε, μέλη της οικογένειας, αν έχουν υπερβεί το 21ο έτος. Ε, επανέφερα παρόλα αυτά τον ορισμό αυτής της οδηγίας μέσα στο δικό μου κείμενο και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε και σε μια συμβαστική λύση και για αυτόν τον ε, ορισμό. Ελπίζω να βρούμε γενικότερα καλές λύσεις ε, και για τους ε, αστέγους και για τους απάτριδες. Όχι αστέγους, απάτριδες εννοούσε η ομιλήτρια και για τους πρόσφυγες. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στις 19 ε, Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενθαρρυντική ήταν η επιστροφή όλων μετά το θέρος.